Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσω τον πρόεδρό μας, Γέρζι Μπούζεκ. Καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή αυτή. Γνωρίζω πόσο ε, μεγάλες δεσμεύσεις έχετε αναλάβει και για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος εδώ και χρόνια. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά. Χαιρετίζω και τον Γενικό Γραμματέα Κλάους Βέλε, ο οποίος επίσης ασχολείται με αφοσίωση με τα θέματα αυτά. Χαιρετίζω και τον Αντιπρόεδρο για περιβαλλοντικά θέματα, την κυρία Ιζαμπέλ Τυρόν. Bonjour Ιζαμπέλ και όλο το προσωπικό και όλους τους συνεργάτες. Υπάρχει μια επισημότητα σήμερα στην τελετή, θα πρέπει να υπογραφεί η δήλωση «Ήμας», το που είναι το πρόγραμμα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς δραστηριοποιούμε υπέρ των περιβαλλοντικών προτύπων και στόχων εδώ και χρόνια και ζητούμε από τους πολίτες και άλλους δρόντες στην κοινωνία να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες. Πολλές. Γι' αυτό είναι σωστό και σημαντικό να δείξουμε και εμείς ότι μπορούμε να αποτελέσουμε πρότυπο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλά. Ε, ο κανονισμός έμας υπάρχει από το 2004 το αναθεωρήθηκε το 2009 και θα ε, προβλέψαμε μια συζήτηση και μετά τη υπογραφή του εγγράφου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, υπάρχουν 27 εθνικά κοινοβούλια και νομίζω ότι είναι σημαντικό το έμας να βγει από το κτίριο αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να φτάσει μέχρι τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, ίσως ε, καλό θα ήταν αυτό να δούμε εάν υπάρχει τέτοια προοπτική καλή συνεργασίας. Ευχαριστώ, σας δίνω το λόγο για την ε, ομιλία σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ακόμα μια φορά βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής ΕΜΒΗ, της Επιτροπής Περιβάλλοντος Άλλους 16 ε, μήνες ε, θα κάθουμε στο θόκο του Προέδρου και μετά θα επανέλθω στην Επιτροπή αυτή. Σήμερα η υπογραφή της ε, δέσμευσης αυτή στα πλαίσια του ΕΜΑΣ είναι πολύ σημαντική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητούσε τα πράσινα θέματα εντό αγωγικών από την αρχή που ιδρύθηκε δηλαδή από τότε που άρχισε να εκλέγεται άμεσα και δημοκρατικά, το 1979. Και ήταν πάντα σημαντικό θέμα. Και από το 1979 έχουμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις για τα περιβαλλοντικά ή πράσινα θέματα. Υπάρχει πολιτική γνώση και πραγματογνωμοσύνη μοναδική σε αυτό το κοινοβούλιο Επομένως, οι ιδέες μας στα πλαίσια του εμάς ε, πρέπει να εξαπλωθούν και να φτάσουν και στα εθνικά κοινοβούλια και αυτή η ιδέα είναι πολύ καλή. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις μας και το βάρος που ασκούμε στο περιβάλλον. Μιλάμε για 17% μείωση του διοξύντου του άνθρακα τα τελευταία έξι χρόνια. Υποσχεθήκαμε επίση ότι θα φτάσουμε το 30% μέχρι το 2020. Ίσως και νωρίτερα. Η... Το ηλεκτρικό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση χαρτιού είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά δημιουργούν αυτό το 17% της μείωσης διοξείδιο του άνθρακα. Την περασμένη εβδομάδα εκδόθηκε μία μελέτη τόσο ώστε να υπάρχει ένα γενικό σχήμα για την αντιστάθμιση των εκπομπών του διοξύδιου του άνθρακα, ένα γενικό πρόγραμμα. Υπάρχει βέβαια και η ατομική ευθύνη του καθενός για να αντισταθμίσει ο καθένας μας τις εκπομπές του στα πλαίσια των ταξιδιών κάνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν συζητούμε για το περιβάλλον, θα πρέπει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προετοιμαστούμε εκ των προτέρων. Και ακριβώς γι' αυτό συναντιόμαστε σήμερα και υπογράφουμε επίσημα τη συμφωνία εμάς. Το πρόγραμμα αυτό οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου για το περιβάλλον. Ενώπιόν μας είναι η συνάντηση του Κανκούν είναι σημαντικό και για την Επιτροπή αυτή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να είμαστε ηγέτε, θέλουμε ακόμα να, είμαστε, να παίξουμε ηγετικό ρόλο και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά στο Κανκούν. Φίλοι, θέλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσαμε δεν πετύχαμε μάλλον την συμφωνία μετά το Κιώτο όπως τη θέλαμε. Αλλά συγκεντρωνόμαστε τώρα σε τρία βασικά σημεία για να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρώτον, το πρόβλημα της ε, καταστροφής των δασών. Πώς θα σταματήσουμε την αποψήλωση των δασών. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, τεχνολογίες. Όλα όσα συνδέονται με τις τεχνολογίες. Ξέρουμε εδώ στην Επιτροπή ΕΜΒΗ, στην Επιτροπή ΉΤΡΕ ότι χωρί νέε τεχνολογίε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά, ότι χωρί νέε τεχνολογίε δεν μπορούμε χωρίς τεχνολογίες να σταματήσουμε την αλλαγή του κλίματος. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προωθήσουμε και τη μεταφορά τεχνολογίας και προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ε, ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα. Μια, ένα τελευταίο σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση είναι η προσαρμογή και ο μετριασμός των επιπτώσεων στο κλίμα και το σχετικό ταμείο. Ξεκίνησαμε πριν από δύο χρόνια. Ε, στην Κοπεχάη πριν από ένα χρόνο βελτιώθηκαν η χρηματοδότηση. Αλλά το να εξοικονομηθούν, το να βρεθούν αυτά τα χρήματα για τις αντισώμενες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, να πετύχουμε μια αύξηση του 3% και να ετοιμάσουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις για το Johannesburg. Όλα αυτά μπορούμε να τα καταφέρουμε και να τα συζητήσουμε στο Cancun. Αυτά έχω να σας πω από τις επαφές που είχαμε διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες και άλλους ηγέτες. 3% είναι η αύξηση χρηματοδότηση. Ε, αυτό επιδιώκουμε να επιτύχουμε στο Κανκούν. Θα ήταν καλά αν το καταφέρναμε. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα συζητήσω μαζί σας τα θέματα που θα θέσω εγώ στο Κανκούν. Θα πάω λοιπόν στο Μεξικό με κάποιους συναδέλφους από το προσωπικό μου γραφείο ε, θα κάτσω μόνο μία μέρα. Δεν θα παραστώ στην ε, διάσκεψη. Ήμουνα στο Ποσνάν, στη Κοπεχάγη. Πριν από τέσσερις μέρες ε, ήμουν στο Ναϊρόμπι. Έχω κάποια εμπειρία. Δηλαδή, Καλύτερα είναι να μην παραστώ στη διάσκεψη. Αλλά το θέμα είναι ακόμα ανοιχτό. Ε, άρχισα πριν από λίγε μέρε να το συζητάω, αυτή την ιδέα δηλαδή, με τον Γιώργο με τον πρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Φυσικά χρειαστεί, μπορώ και να παραστώ, αλλά υπάρχουν και λόγοι του οποίου καλό θα ήταν να μην παραστώ. Αυτά. Uh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε τη δέσμευσή σας ε, υπέρ ε, της διατήρησης του κλίματος. Στο Κανκούν θα ξεκολουθήσουμε να έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες, θα προετοιμάσουμε και ένα ψήσμα για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου, θα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και στην Ολομέλεια σε κάποιο μεταγενέστερο χρονικό σημείο και η φιλοδοξία μας βέβαια είναι να έχουμε μια συνολική συμφωνία για την προστασία του κλίματος. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτό το οποίο θα διαπραγματευτούμε στο Κανκούν είναι κάποιες πτυχές για την επίτευξη αυτής της συνολικής παγκόσμιας συμφωνίας. Και ίσως επανέλθουμε αργότερα στο Ιωάννεσμπουργκ και να καταλήξουμε δηλαδή σε μια συνεκτική, μια πλήρη συμφωνία. Πάντως για όλα αυτά είναι απαραίτητο ήδη κάποια τμήματα της συμφωνίας να τα έχουμε ήδη πετύχει στο Κανκούν. Μακάρι να έλθετε εκεί, να είστε μαζί μας. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, έχετε να διεκπαιρεώσετε διαπραγματεύσεις και σε άλλους τομείς. Πάντως ε, θα είστε ψυχήτε και πνεύματι, αν όχι σώματι, μαζί μας στο Μεξικό, στο Κανκούν. Σας ευχαριστώ πολύ και να δώσω τώρα το λόγο στην Αντιπρόεδρό μας, την Ιζαμπέλ Ντιγόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε από τη δική μου πλευρά, εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα ΕΜΑΣ, ε, με το οποίο είμαι επιφορτισμένη ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ελπίζω να, ως αντιπρόεδρος να είναι το αντίθετο του greenwashing, να μην μετριαστούν δηλαδή τα οικολογικά θέματα και σημασία τους ε, στο Κοινοβούλιο. Ε, δεν είμαστε μόνο αυτοί που νομοθετούμε, είμαστε αυτοί που δίνουμε και το παράδειγμα και το καλό παράδειγμα. Για να το πράξουμε αυτό όμως θα πρέπει τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας να είναι πραγματικά εργαλεία. Δηλαδή, τι νόημα έχει να αγοράζουμε, να χρησιμοποιούμε λιγότερο ρηπογόνα οχήματα εάν ε, τα κινούμε περισσότερο. Γιατί ξέρετε ότι τότε θα έχουμε μεγαλύτερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί να χρησιμοποιούμε πιο καλέ ή καθαρέ πηγέ ενέργεια, αν χρησιμοποιούμε περισσότερη, αν καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια. Το έμας λοιπόν είναι κάτι πολύ καλό για όλου μα εδώ για να ε, κάνουμε μια πραγματικά γνήσια προσπάθεια πολέμηση τη αλλαγή του κλίματο για να τα καταφέρουμε καλύτερα, να καταφέρουμε επίση περισσότερα από ό,τι έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό επίση καλό είναι και εμεί ω βουλευτέ να κινητοποιηθούμε, αλλά να κινητοποιηθεί το σύνολο του προσωπικού, το σύνολο θεσμικού οργάνου και Όλοι πρέπει να συμμετέχουν ε, στην υλοποίηση του αίμα σε καθημερινή βάση για να το πετύχουμε. Αν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ πιο αξιόπιστοι, θα έλεγα 100 φορέ πιο αξιόπιστοι και προ τα έξω, όταν προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την πολιτική μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα το πετύχουμε αυτό αν δείξουμε και εμεί ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι ένα κοινοβούλιο που δεν εκπέμπει καθόλου ε, διοξίδιο του άνθρακα, μηδενικέ εκπομπέ, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε να εξοικονομήσουμε τουλάχιστον. Και εμεί ε, στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνουμε προσπάθειες και αν δείξουμε ότι με σοβαρή οικολογική προσπάθεια και με αποφασιστικότητα μειώσουμε και το λειτουργικό μας κόστος, το κόστος λειτουργία, θα έχουμε κερδίσει και από περιβαλλοντική πλευράς και από πλευρά ε, τη υπευθυνότητα που δείχνει το Κοινοβούλιο στη χρήση των δημοσίων κονδυλίων που έχει στη διάθεσή του. Θα υπογράψουμε λοιπόν και για ε, το χάρτη της επόμενης χρονιάς, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε την πολιτική αυτή. Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος άλλωστε έχουν και μία παραπάνω ευθύνη, ίσως από όλους εμάς, γιατί φυσικά δεν μπορεί να νομοθετεί κάποιος από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να μην ε, κάνει αυτό το οποίο οφείλει και μπορεί να πράξει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο λοιπόν αυτό το σύστημα. Σίγουρα μπορούμε ως κοινοβούλιο να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα στον τομέα του περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ακούσουμε τώρα παρεμβάσεις από τις ε, πολιτικές ομάδες. Γνωρίζω Υπάρχουν περιορισμοί στο έργο μας και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Μετακινούμαστε συνεχώς από τη μία πόλη στην άλλη. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό τώρα ούτε σήμερα ούτε σε αυτή την Επιτροπή. Ας ακούσουμε όμως κάποιες παρεμβάσεις. Λίντα Μακάβαν η συγγήτρια για τον κανονισμό εμάς, ίσως θα ήταν καλό να λάβει πρώτη το λόγο για δύο-τρία λεπτά. you, need... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζομαι τρία λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρό μας όμως, γιατί ξέρω πόσο σοβαρά προσεγγίζει τα θέματα της κλιματικής αλλαγής εργάστηκε και στην ε, Κοπενχάγη και στο Μπαλί και αλλού για πρόοδο. Εμείς γνωρίζουμε ότι πολλά μπορεί να γίνουν καλύτερα και στα κτίρια μας για εξοικονόμηση ενέργειας. Γι' αυτό το έμας είναι τόσο σημαντικό. Όταν ε, συμφωνήσαμε πέρσι για τις αλλαγές στο ΙΜΑΣ, θέλαμε να δείξουμε ότι πρώτα θα νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας και είναι πάρα πολύ καλά τα νέα για την αντιστάθμιση του άνθρακα και η ανακύκλωση μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο. Αυτό πολλές φορές το έχουμε πει και πολλά παράπονα έχουν γίνει. Τα πλαστικά μπουκάλια από τα γραφεία πού πάνε, στο Στρασβούργο είναι χωριστά. Ένα απλό παράδειγμα σας δίνω, δεν είναι το ίσως τόσο γλαφυρό. Αλλά υπάρχουν στο Στρασβούργο διαφορετικοί κάδοι για διαφορετικά πράγματα. Αλλά μετά έρχονται για τη συλλογή και τα βάζουν στον ίδιο σάκο. Οπότε δεν γίνεται διαλογή για ανακύκλωση στο Στρασβούργο, ίσως ούτε και στις Βρυξέλλες. Πολλά μπορούν να γίνουν όμως. Και βέβαια θέλουμε το είμαστε να εφαρμοστεί σε πολλούς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι είχαμε ένα σύστημα απλοποίησης, το οποίο θεσπίσαμε για να, να το κάνουμε αυτό. Βέβαια και στο, έχω εκεί τρει έδρε στο Κοινοβούλιο, Βρυξέλλε, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, διαφορετικέ χώρε, εφαρμόζουν διαφορετικά τον νόμο. Άρα δυσκολεύεται και το Κοινοβούλιο να εφαρμόσει το «ή» μα έτσι. Γίνεται σαφέ ε, ότι δεν μπορούμε να, αν εμεί δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, άλλε εταιρείε που έχουν διαφορετικέ έδρε και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικού τόπου, θα έχουν ε, προβλήματα. Ε, Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε το παράδειγμα και πολλές εταιρείες να ακολουθήσουν περιορίζοντας το αποτύπωμα του άνθρακα και φροντίζοντας το περιβάλλον εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, προσβλέπουμε στην αλλαγή που θα λάβει γύρω μας και θέλουμε να συμμετάσχουμε στο «Ήμας». Ευχαριστώ. Ο Ρίχαρντ Ζέμπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που έχουμε τον Πρόεδρο Μπούζεκ και τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Καλώς ήρθατε. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το ε, εθέλοντικό ε, πρόγραμμα που επιβάλλει το Κοινοβούλιο. Βέβαια θα πρέπει να ε, δούμε τι μπορούμε να, να βελτιώσουμε και σε νομικό επίπεδο για το Κανκούν ε, είναι καλό να συμμετάσχετε, ιδιαίτερα τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι σημαντικό στο Κοινοβούλιο να δώσουμε σαφές μήνυμα. Ε, βεβαίως, ε, ε, ο Γιώ είναι εξαιρετικός, δεν θέλω να τον υποτιμήσω προς Θεού, αλλά η παρουσία του Γέρση Μπούζεκ θα τόνιζε τη σημασία που προσδίδει στη διάσκεψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την υπόθεση αυτή του ΕΜΑΣ θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες λεπτομέρειες. Ανέφερε ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος ότι πρέπει να δίνουμε καλά παραδείγματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω να δείτε τι γίνεται με τον διαγωνισμό ε, για την υπηρεσία των οδηγών. Ε, είναι σημαντικό να οργανώσουμε καλύτερα την υπηρεσία των οχημάτων μας. Μπορούμε με εξορθολογισμό να εξοικονομήσουμε 10% μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι οικιστικό το μέτρο. Ε, μιλήσαμε για τα... και ψηφίσαμε την έκθεση για τα ε, πρότυπα για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, γιατί όχι και εμείς τώρα, για το κάπνισμα έχουμε ε, παντού ε, τις πινακίδες για, το, για να μην καπνίζομαι. Θα πρέπει να τηρούμε και εμείς τους κανόνες που θεσπίζουμε για τους άλλους. Θα πρέπει δηλαδή και εδώ στο Κοινοβούλιο να μην καπνίζομαι, αλλιώς είμαστε αναξιόπιστοι. Και τα ύδατα, το αγαπημένο μου θέμα. Δεν έχω την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο αυτό ε, λειτουργεί με τρόπο ορθολογικό εις ό,τι αφορά την εξοικονόμηση. Βεβαίω, υπάρχουν, ε, υπάρχει ε, ποσότητα υδάτων, αλλά όμως έχουμε στην ημερήσια διάταξη την απόδοση κτηρίων ως προς την κατανάλωση ύδατος. Και γι' αυτό και εδώ θα πρέπει να δώσουμε πρώτη το παράδειγμα. Ναι, στο Στρασβούργο ε, είναι πάρα πολύ καλό το σύστημα ε, τον, ε, με τις βρύσεις που έχουμε στο Στρασβούργο γιατί είναι λίγο το νερό που καταναλώνουν. Chris Davis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω όπως και οι συναδελφοί μου τις ρυθμίσεις αυτές. Τα μέλη της Επιτροπής μας θα ενθαρρύνουν μια παρουσίαση του έμας, αν όχι στο, στην Επιτροπή, σε ένα σεμινάριο για μέλη της Επιτροπής μας και άλλους. Να πάρουμε δηλαδή, να, να παίξουμε έναν ηγετικό ρόλο και να ενθαρρύνουμε ε, τα πράγματα και να δώσουμε και πολιτική στήριξη όπου χρειάζεται. Ε, σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, ή ε, οπουδήποτε ε, κατασκευάζονται μηχανήματα, μηχανές, ε, η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία τους είναι η διαχείριση μέσα από τη μέτρηση. Όταν πρόκειται για εκπομπές, χρήση ύδατος, κατανάλωση ενέργειας, χρήση πόρων, απορρίμματα, όλα αυτά σε μια αυτοκίνητο βιομηχανία ρυθμίζονται και ενημερώνεται ο κόσμος που δουλεύει εκεί στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Δηλαδή αυτά κάνουμε, αυτό είναι ο στόχος κλπ. Ε, ε, Πού λοιπόν θα ήταν ένας κατάλληλος χώρος να αναρτήσουμε και εμείς τέτοιου είδους πινακίδες και οι επισκέπτες να ε, μπορούν να βλέπουν και να τους δείχνουμε τα στοιχεία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα και για το Κοινοβούλιο και για ε, άλλα εθνικά κοινοβούλια και για άλλα θεσμικά όργανα. Κάρλος Σλούκα, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πρόσφατα με διορίσανε υπεύθυνο για το ΕΜΑ σε αυτή την Επιτροπή. Σας καλωσορίζω κύριε Μπούζεκ ε, στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι Υπάρχουν πολλές ελλείψεις ακόμα. Πριν από 10 χρόνια αποφασίσαμε ότι το 5% της ενέργειάς μας ε, θα παράγεται από εμά του ίδιους. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά τίποτα τέτοιο στο Κοινοβούλιο. Πού είναι αυτό το 5% που το αποφασίσαμε, γιατί δεν το υλοποιούμε. Και, για και γιατί επίσης ε, χρησιμοποιούμε αυτά τα χαρτιά, θα μπορούσαν να είναι πιο λεπτά τα χαρτιά. Και επίσης γιατί χρησιμοποιούμε τα πλαστικά μπουκάλια. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε πλαστικά μπουκάλια. Ή αυτές οι, αυτοί οι λαμπτήρες. Νομίζω ότι είναι ακριβό το να σκαρφαλώνουμε και να τις αλλάζουμε. Ε, υπάρχουν... έχουμε αποφασίσει στην Ευρώπη να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε λαμπτήρες με, με υδράργυρο. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, λαμπτήρες LED. Είναι πιο ακριβές ίσως, αλλά νομίζω ότι κρατάνε περισσότερο και αξίζει τον κόπο. Επίσης, οι υπολογιστές. Κάθε χρόνο έχω καινούριο κομπιούτερ, είτε εδώ είτε στο Στρασβούργο. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, αυτή την αλλαγή. Είναι θέμα διαχείρισης. Στη Σουηδία, στις ε, τοπικές αυτοδιοικήσεις, Ε, είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Εδώ, ας πούμε, ε, έχουμε οπτικές ίνες, έχουμε όλα τα προγράμματα, έχουμε κεντρικούς υπολογιστές και κάθε υπολογιστής που χρησιμοποιούμε στο γραφείο μας είναι απλό τερματικό. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους παλιούς ε, κομπιούτερ για 10 χρόνια. Δεν ξεπερνιόνται γιατί ο επεξεργαστής τους κρατάει. Και ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αλλάζει κεντρικά στο κοινοβούλιο. Ε, επομένως, ε, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε εμεί κάθε φορά τον ατομικό μα υπολογιστή. Έτσι κερδίζουμε χρόνο, ε, εξοικονομούμε υπολογιστέ, εξοικονομούμε ενέργεια, χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια. Αυτά τα απλά πράγματα πρέπει να τα συζητάμε περισσότερο. Ή τα αυτοκίνητα. Γιατί να μην έχουμε την επιλογή να έχουμε πιο μικρά αυτοκίνητα που είναι και πιο εύχριστα για του οδηγού. Γιατί όχι. Και γιατί να μην παίρνουμε το ποδήλατο στο σπίτι και να ερχόμαστε από το σπίτι με αυτό. Γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μόνο μέσα στη μέρα δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα παίρνουμε ε, στο σπίτι και να ερχόμαστε στη δουλειά ε, με το ποδήλατο. Αυτές είναι μικρές ε, συστάσεις που θα κάνω από την καθημερινή μου ζωή ως ευρωβουλευτή. Όλοι έχουμε τέτοιε ιδέες, ας τις ακούσουμε και ας τις υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολλές ιδέες ακούστηκαν από την Επιτροπή. Ο Chris Davis είπε να κάνουμε ένα ατελείο, ένα εργαστήρι για το εμάς, για να επεξεργαστούμε, να συζητήσουμε αν θέλετε όλες αυτές τις ιδέες. Έχετε το λόγο πριν περάσουμε στην επίσημη υπογραφή του εγγράφου. Ωραίες είναι αυτές οι ιδέες που προτείνει ο τελείο Για τους λαμπτήρες ας πούμε και το ηλεκτρικό ρεύμα και το φωτισμό. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τη διοίκησή μας να μας πει τι πρέπει να τι μπορούμε να κάνουμε σε 10 σημεία, στα πλαίσια του εμάς. Και μία από τις ιδέες είναι να αλλάξουμε όλους τους λαπτήρες του χρόνου. Θα κοστίσει ένα με 2 εκατομμύρια. Αλλά θα, αποδώσουν, θα αποδώσει αυτή η δαπάνη σε 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια αυτά τα λεφτά θα είναι σαν να τα παίρνουμε πίσω. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, δεν είναι λίγο. Επίση θα ετοιμάσουμε και ένα κοιτίο για ιδέες. Αν Έχουμε, έχετε βέβαια εσεί ε, ιδέε με το Γενικό Γραμματέα, ε, συγγνώμη, συναντήσει με το Γενικό Γραμματέα, τότε δεν χρειάζεται αυτό κουτί. Γιατί τότε συζητάτε αυτά τα θέματα. Αλλά όλα αυτά τα λέω γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί γιατί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεισφέρουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ηγέτε, να παίξουμε ηγετικό ρόλο και στην Ευρώπη και στον κόσμο, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι το μήνυμα, λέει ο Πρόεδρο. ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που ήρθατε. Η τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εδώ. Και έτσι υπάρχει κάλυψη από τα ΜΜΕ. Ας περάσουμε στην υπογραφή του κειμένου και αδεσμευτούμε για την δεύτερη περίοδο λειτουργίας του ΕΜΑΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Μετά τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου έχω την τιμή να καλωσορίσω την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Δαμανάκη. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος η πρώτη σας επιτροπή είναι η Επιτροπή Αλίας βέβαια, δεν συζητείτε και αυτή η συζήτηση όμως ζητήθηκε από τα μέλη και είπα μη φοβάστε ε, πολιτική αλίας, δεν θέλουμε να κάνουμε υπέρβαση αρμοδιοτήτων εδώ, αλλά το θαλάσσιο περιβάλλον μας αφορά και μας τόσο πολύ, αφορά τόσο πολύ τη δουλειά μας, που είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε για τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνεται για μια βιώσιμη και αηφόρο πολιτική σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Ιδιαίτερα, ειδικότερα σήμερα το πρωί, περάσαμε ένα, εγκρίναμε ένα ψήφισμα για τις εξορίξεις πετρελαίου στη θάλασσα και τι μπορεί ιδιαίτερα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικά της ύδατα. Θυμάμαι την εξαιρετική σας ομιλία στο Στρασβούργο πριν από τις θερινές διακοπές ακόμα επί του θέματος αυτού. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν σαφέστατη, ήταν συνεπής ε, σχετικά με τις υψηλές ε, προδιαγραφές που θέτομε σε όσους δραστηριοποιούνται σε τέτοια κλίμακα αξιοποιώντας τους πόρους. Αλληλεία, περιβάλλον, ένα περίπλοκο θέμα το οποίο πολλές φορές έχει ταλαιπωρηθεί. Ε, και πάλι ένα θερμό καλώς ήλθατε και σας δίνω το λόγο αμέσως για να μας μιλήσετε για την ανάπτυξη των ιδεών και τα προγράμματά σας για την αλληλεία. Dear Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε Λάινον, αξιότιμοι βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με προσκαλέσατε να έρθω εδώ στην Επιτροπή σας για να συζητήσω μαζί σας την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μας διαφύγει το γεγονός ότι τα ζητήματα τα οποία ασχολούν την Επιτροπή σας ε, σχετίζονται στενά με την αλία. Γι' αυτό λοιπόν και δέχθηκα με μεγάλη χαρά την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ και πραγματικά θα ήθελα να συνεργαστείτε μαζί σας. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα να ασχοληθείτε με τα θέματα που απασχολούν ε, την, ε, ε, το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Γιατί μόνο έτσι θα στηρίξουμε τη βιωσιμότητα και τις προσπάθειες από γίνονται. Για να το πω με άλλα λόγια, για να πετύχουν οι πολιτικές μας θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ ε, του τμήματος της αλίας και του τμήματος του περιβάλλοντος, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε τους κοινούς στόχους και των δύο πολιτικών. Όπως λοιπόν αναφέρατε, ποτέ δεν έκρυψα την επιθυμία μου περιβαλλοντικοί παράγοντες να είναι στο επίκεντρο της μεταρρύθμισής μας. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι χρειάζεται πραγματικά μια προσέγγιση οικοσυστήματος για τη διαχείριση της αλίας. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε την ολοκληρωμένη πολιτική της θάλασσας και τον περιβαλλοντικό πυλώνα, δηλαδή ε, την οδηγία πλαίσιο ε, για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχος μου λοιπόν είναι να διαμορφώσω μια μελλοντική πολιτική η οποία θα συμβάλλει στους στόχους της ε, θαλάσσιας στρατηγικής. Η νέα μας πολιτική δηλαδή πρέπει να επιτύχει και να διατηρήσει ε, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για την πολιτική μα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε η αλληλεία να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε τα αλλιεύματα, τα αποθέματα αλλά και τα ε, θηλαστικά και τα θαλάσσια πτηνά να μπορούν να αναπαράγονται και να αυξάνονται οι πληθυσμοί του. Θα πρέπει λοιπόν η αλίευση να γίνεται σε βιώσιμα επίπεδα και να μην υπάρχουν παρεμπίπτοντα αλλιεύματα μεταξύ αυτών γόνι δηλαδή. Δεν θα πρέπει η αλλίευση λοιπόν να υπονομεύει τους στόχους διατήρησης της βιοποικιλότητας πρέπει να γίνουν σεβαστές και υποχρεώσουμε στο πλαίσιο του Natura 2000. Θα πρέπει επίσης να μειωθεί για να μην να σταματήσει η πρακτική της απόρριψης. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τις απορρίψεις πια. Η κοινή αλληλευτική πολιτική, ως έχει αυτή τη στιγμή, πραγματικά υπολείπεται όλων αυτών των στόχων. Αυτό το καταστήσαμε σαφές ε, στο πλαίσιο του πράσινου βιβλίου. Και συμφώνησαν μαζί μας ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων φορέων, όχι όλοι, πάντως πολλοί. Έχουμε λοιπόν μία υπεραλίευση ε, των αλληλευτικών στόλων. Αυτό είναι μία μόνιμη κατάσταση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κοντόθωρη ε, προσέγγιση. Το έχουμε δει και στις ετήσιες ε, συναντήσεις του Συμβουλίου γιατί γίνεται συζήτηση για μεγαλύτερες ποσοστώσεις. Είναι καταστροφή, πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Το έχω προσπαθήσει και πριν από τη μεταρρύθμιση της πολιτικής το έχω ξαναπεί και σε εσά και θέλω να το επαναλάβω. Θέλουμε την υποστήριξή σας. Μην με παρεξηγήσετε όμως, η αποτυχία αυτής της πολιτικής δεν είναι αποκλειστική υπετιότητα του Συμβουλίου. Φυσικά ε, και είναι υπόλογο και το Συμβούλιο, δεν είναι όμως το μόνο. Πρέπει να πω ότι η προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση δεν δίνει επαρκή ιδιοκτησία και ευθύνη στον ελευτικό κλάδο. Αν πάρετε τα τρία προβλήματα, υπερ, ε, υπερβολικές δυνατότητες, υπεραλίευση, η προσέγγιση top-down από την κορυφή προς τη βάση αν προσθέσετε και την κοτόθωρη πολιτική, καθώ και το γεγονό ότι πολλέ φορέ δεν υπήρξε απαραίτητη πολιτική βούληση για την ε, σωστή εφαρμογή, έχετε και τη συνταγή τη καταστροφή. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Το έχω πει επανειλημμένο, το επαναλαμβάνω και στο σώμα αυτό και αλλού. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Πολύ απλά. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια εκβάθρον μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και πρέπει μια και για πάντα να εγκαταλείψουμε την παλιά πεποίθηση ότι δεν είναι συμβατή η αλληλευτική πολιτική με την περιβαλλοντική πολιτική. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι θα πρέπει να καθιερωθεί η προσέγγιση του οικοσυστήματος πιο άμεσα με τη μεταρρύθμιση της τρέχουσας ε, κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Στο αποτέλεσμα η αλληλευτική πολιτική θα καλύπτει μέτρα όπως προστασία κάποιων ευαίσθητων περιοχών, όπως αυτό που γίνεται η αναπαραγωγή και η επόαση και κάποιες άλλους τομείς. Η νέα πολιτική θα πρέπει να προστατεύει επίσης και μη στοχευμένα είδη όπως είναι τα κοιτοειδή, οι καρχαρίες, τα θαλάσσια πτηνά και θα χρησιμοποιεί κάποια εργαλεία της αλληλευτικής πολιτικής όπως ειδικό σχεδιασμός παραδείγματο χάρη στον τομέα της θαλάσσιας στρατηγικής ούτως ώστε να υπάρχει πλήρη συντονισμός όλων των αλληλευτικών και ναυτιλιακών ε, ζητημάτων για τη θάλασσα και του πόρου τη. Πρέπει επίσης να ενσωματώσουμε καλύτερα τα μέτρα αυτά σε μακροπρόθεσμα σχέδια. Μακροπρόθεσμα σχέδια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόθεσή μου λοιπόν είναι να επεκτείνω τα μακροπρόθεσμα προγράμματα για όλα τα εμπορικό σημαντικά αληφτικά είδη αυτή η αισιόδοξη, αν θέλετε, διάθεση για τους στόχους μας, ε, για την πολιτική, συνοδεύεται όμως και από μια προειδοποίηση και θέλω να είμαι ειλικρινής ε, απέναντί σας. Όλες αυτές οι αγαθές προθέσεις δεν θα παραμείνουν παρά μόνο μια τρύπα στο νερό, εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας. Πρέπει να αποφύγουμε την μικροδιαχείριση σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να εστιάσουμε στα αποτελέσματα, στην ε, στόχοθέτηση και να επιλέξουμε επίσης και τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των πολιτικών μας στα κράτη-μέλη. Αυτό ακριβώς θα πράξουμε. Θέλουμε ένα σύστημα όπου η ελληνική βιομηχανία αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετέχουν με το σωστό τρόπο και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τις απαραίτητες ευθύνες. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίσουμε για μια πραγματική βελτίωση ό,τι αφορά τη συμμόρφωση. Εξού και επαναλαμβάνω, αυτό που θέλω είναι πιο οικολογική, πιο απλή και πιο αποκεντρωμένη αλληλευτική πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημά μας και αυτό είναι και ο στόχο μα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες όταν θα φτάσουμε στον ώρα του καθορισμού των βασικών στόχων. Αν έχουμε στόχους ε, που είναι αντιπαρατηθέμενοι ένας προς τον άλλον, ε, θα μας οδηγήσουν πάλι σε κάποιες κοντόφερες προσεγγίσεις. Για μένα προσωπικά η κοινωνική πολιτική της πολιτικής είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με τις άλλες, σας, γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Αλλά, αλλά, πρέπει να πω ξεκάθαρα εδώ, ότι πρέπει το ίδιο ξεκάθαρο να είναι σε όλους τους άλλους. Ότι δηλαδή αν δεν έχουμε υγιή ε, αλλιευτικά αποθέματα και ανθούντα οικοσυστήματα, δεν θα μπορέσει να υπάρχει κάποια κοινωνική τάση. Η βιωσιμότητα είναι ο μόνος ε, τρόπος για να έχουμε άνθηση της αλληλευτικής κοινότητας στην Ευρώπη. Είναι και καλύτερη πολιτική για την εξασφάλιση των αλλιέων και των οικογενειών τους. Η βιωσιμότητα λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα. Και Έρχομαι λοιπόν με την κοινωνική διάσταση στο ζήτημα της μικρής κλίμακας αλίας. Πρόκειται για αλία η οποία πολλές φορές ε, σε ζωτικό βαθμό μάλιστα συμβάλλει ε, στην, ε, στον κοινωνικό ιστό και στην οικονομική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων που είναι πάρα πολύ σημαντικές όπως γνωρίζετε ήδη πολύ καλά. Επομένως τα πλοία τα οποία ασχολούνται με, με την μικρή κλίμακα αλίας πολλές φορές προκαλούν λιγότερη ζημία στο περιβάλλον και πολλές φορές είναι πιο επιλεκτικά ε, στις αλληλευτικές δραστηριότητες ε, από ότι άλλα τμήματα του αλληλευτικού στόλου. Γι' αυτό λοιπόν για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας και το στόλο αυτό στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών μας. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να τονίσω το εξή. Η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν αφορά μόνο έναν σχετικά μικρό τομέα, τον τομέα της αλλήλευσης, καλύπτει και την κοινή αγορά των αλληλευτικών προϊόντων, εκ των οποίων πάνω από το 50% προέρχεται από εισαγωγέ. Το 50% των ψαριών που καταναλώνουμε προέρχεται από εισαγωγέ. Επομένω, δικό μου καθήκον και δεδηλωμένο στόχος μου είναι να προωθήσω τη βιώσιμη αλία πέραν των κοινοτικών υδάτων μέσω του πολυμερούς πλαισίου, μέσω των περιφερειακών οργανώσεων ε, διαχείρισης αλίας και μέσω διμερών συμφωνιών. Θα εξασφαλίσω λοιπόν τη συμπερίληψη της ε, εξωτερικής αυτής διάστασης στην ε, ημερήσια διάταξη της μεταρρύθμισης. Και όπως ίσως γνωρίζετε, Προτίθεμαι επίσης να προτείνω και μια θεμελιώδη αναβάθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους βασικούς στόχους και αρχές ε, της ε, μεταρρυθμισμένης κοινή ε, αλλιευτικής πολιτικής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε στους καταναλωτές ότι τα ψάρια που αγοράζουν προέρχονται από υγιείς και βιώσιμε πηγέ και πρέπει να βρούμε πραγματικά τον τρόπο και τη σωστή κατάλληλη σήμανση, επισήμανσης στι ετικέτες για το τέλος έχω αφήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και πρόκειται συγκεκριμένα για τη συναπόφαση. Η μεταρρύθμιση αυτή θα είναι η πρώτη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα αποφασιστεί από κοινού, από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Επομένως, προσκαλώντας με σήμερα εδώ, έχετε ήδη δείξει ε, ότι συμμετέχετε ενεργά στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας όταν φτάσουμε στη συζήτηση και την ε, διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιτευξη μια πραγματικής μεταρρύθμισης. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που ακούγονται και υποστηρίζουν ότι η μεταρρύθμιση μπορεί να γίνει με μικρές παρεμβάσεις ε, από εδώ και από εκεί. Τις ακούω και θα τις ακούσω αυτές τις φωνές. Είμαι ωστόσο πεπισμένη ότι δεν αρκεί κάτι τέτοιο να σφίξουμε δύο-τρεις βίδες από εδώ δηλαδή και να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε σημαντικές προκλήσεις οι ιδέες που ανταλλάσσουμε σήμερα θα τροφοδοτήσουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις που έχουμε για το πώς θα προχωρήσουμε με τη μεταρρύθμιση μας. Σας προσκαλώ θερμά λοιπόν να συνεχίσετε να συμμετέχετε ενεργά στη διαδικασία μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και προσβλέπω στην ε, συνεργασία με το Κοινοβούλιο σας κατά τους επόμενους μήνες και έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Κυρία Επίτροπε Δαμανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, σαφέστατη παρουσίαση της πολιτικής σας. Δεν μας απαγοητεύσατε. Πρόκειται για μια συνέχεια ε, προηγουμένων ομιλιών σας. Έχουμε αυτή την ε, οικολογική προσέγγιση στην αλληλεία που θέλουμε να την υποστηρίξουμε. Την υποστήριξη τη θέλετε και εσείς. Άλλωστε, Αρχίζουμε τη συζήτηση. Οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για τις ε, ε, παρεμβάσεις της. Ε, είναι πολύ σημαντικό να την υποστηρίξουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αηφορία Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη υπεραλίευση σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να καταφέρουμε στην Ευρώπη να αποκαταστήσουμε κάποια ισορροπία. Στην Ισλανδία εντυπωσιάστηκα με τα αποτελέσματα που έχουν εκεί και πώς ε, βελτίωσαν την πολιτική αλίας τους. Νομίζω ότι χρειάζεται απλή πολιτική με σκληρές κυρώσεις και απλό σύστημα. Ο έλεγχος βέβαια είναι δύσκολος όπως και η επαλήθευση. Και εδώ θα πρέπει να απλουστεύσουμε, να βελτιώσουμε τη δυνατότητα ελέγχου, αλλά μετά να προβλέπονται ε, αυστηρές κυρώσεις. Και τότε θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ε, διασφάλιση της αηφορίας στην αλληλεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Natura 2000 και την βιοπικιλότητα, ξέρουμε όλοι ότι τώρα έχουμε μεγάλη υποβάθμιση της βιοπικιλότητας. 10% των περιοχών της Natura 2000 είναι θαλάσσιες περιοχές, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα να προτείνετε περιοχές Natura 2000, αλλά οπωσδήποτε καλό θα είναι να υποστηρίξετε κι εσείς για τον καλύτερο ορισμό των προστατευομένων περιοχών θα ήταν ε, ευπρόσδεκτη δηλαδή μια δική σας παρέμβαση σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ρίχαρτ Ζέμπερ. Ο Κρήτον Αρσένης. Ε, να σας καλωσορίσω Επίτροπε. Ε, πραγματικά οι κατευθύνσεις που παρουσιάσατε μας βρίσκουν και με βρίσκουν προσωπικά σύμφωνο. Ε, θα ήθελα να, να ρωτήσω δύο-τρεις εξειδικευμένες ερωτήσεις Πρώτο, ε, βλέπουμε σε πολλά κείμενα τη Επιτροπή να εξετάζονται πολλά εναλλακτικά σενάρια. Παραδείγματο χάρη στην περίπτωση του τόνου. Ε, βλέπουμε να εξετάζονται σενάρια, τα οικονομικο-κοινωνικέ επιπτώσει, αν ενταχθεί ε, στην, ε, στο Appendix 1, Appendix 2, του Άντε κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε το σενάριο τη κατάρρευση να εξετάζεται. Ποιε είναι οι επιπτώσει. Αν αυτό σκέφτεστε να αλλάξει. Και δεδομένου ότι ο τόνο απειλείται από κατάρρευση, ε, αν αυτό που αναφέρεται για απαγόρευση αλίας σε περιοχές εοδοκία, αν το σκέφτεστε σαν μέτρο πιθανό για την περίπτωση του τόνου. Ε, τέλος, ε, και περιμένουμε με, μεγάλη, με μεγάλο ενδιαφέρον την εκτίμηση επιπτώσεων της ε, κοινής αλληλευτικής πολιτικής που έχει ανακοινωθεί για, τον, ε, για το φθινόπωρο ε, και αν στα πλαίσια της ε, νέας αλληλευτικής πολιτικής και στα πλαίσια των συμφωνιών που θα υπάρχουν από εδώ και εμπρός ε, να, να υιοθετήσετε αυτό που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο σε πρόσφατο ψήφισμα, που είναι δηλαδή ε, να γίνονται αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες μόνο όταν είναι επιστοποιημένο ότι υπάρχει επάρκεια για τους αλείς εκεί πέρα, για τους τοπικούς πληθυσμούς των φτωχών χωρών και την ίδια στιγμή ε, υπάρχει βιολογικό πλεόνασμα των αλληλευμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Chris Davis. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Τα καλωσορίζουμε. Το έχω ξαναπεί ότι θεωρώ τη δουλειά που κάνετε από τις πιο σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν κοιτάξουμε την, τη σημερινή στιγμή μετά από χρόνια και αυτά που πέτυχε η Ευρώπη, εάν καταφέρετε με τη μεταρρύθμιση την αλληλευτική να βάλετε κάποια ψάρια στις θάλασσές μας, να αυξηθούν τα ψάρια στις θάλασσές μας, θα είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα αυτό. Ένα-δύο ερωτήματα. Ίσως τα απαντήσατε. Αλλά ακούω διάφορες φήμες ότι μειώνετε τις φιλοδοξία σας. Γιατί υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, λέει. Εσείς ξεκαθαρίσατε όταν μιλήσατε ότι θέλετε ε, βαθιά και πλατιά μεταρρύθμιση. Οι φήμε όμως που ακούγονται είναι ότι υποκύπτεται στις πολιτικές πιέσεις, εν πάση στην πολιτική πραγματικότητα. Ίσως θα θέλετε να το σχολιάσετε αυτό το σημείο. Δεύτερον, για τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Η κοινή αλληλευτική πολιτική αυτό που θέλει να πετύχει είναι να κρατήσει σταθερά τα αποθέματα και σε μερικέ περιπτώσει να τα βοηθήσει να ανακτήσουν. Αλλά τα επίπεδά του είναι πολύ κάτω από το δυναμικό των θαλασσών μας. Και είναι ευάλωτη η κατάστασή τους. Για να φτάσουμε σε καλύτερη κατάσταση, για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή βιώσιμη απόδοση, απόδοση περισσότερα ψάρια στις θάλασσες, μεγαλύτερη βιοπικιλότητα, καλύτερη κατάσταση για τους ε, ψαράδες, όπου να μειώσουμε την αλίευσή μας. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια δύσκολη περίοδος, όπου θα μειώσουμε την αλληλευτική μας προσπάθεια, ούτως ώστε να πετύχουμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Το πολιτικό ερώτημα που τίθεται είναι, εσείς μιλήσατε στο Συμβούλιο, τι πολιτική στήριξη έχετε για τις απαραίτητες αλλαγές. Τι υπάρχει καταρχάς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι πολιτική στήριξη. Σας υποστηρίζει ο Πρόεδρος, αναγνωρίζει το σημαντικό σας καθήκον και μέσα στο Συμβούλιο. Δεύτερον, υπάρχουν φωνές που αναγνωρίζουν την ανάγκη να κάνουμε ουσιαστικές μακρόπνοες αλλαγές ή θα σας καθυστερήσουν και το Δεκέμβριο και τα επόμενα χρόνια με αυτές τις κοντόθωρες απόψεις και πολιτικές τους. Tough Δύσκολες ερωτήσεις. Για να δούμε και τις απαντήσεις. Σαντρίν Μπελιέ. Ευχαριστώ. Κυρία Δαμανάκη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί είσαστε παρούσα στην Επιτροπή μας σήμερα και να σε ευχαριστήσω επίσης για την θαραλέα σας θέση τον Ιούνιο για τις ποσοστώσεις για τον ερυθρό τόνο. Θέλω πραγματικά να επωφεληθώ από τη σημερινή ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας, για το θάρρος σας στον τομέα των ποσοστώσεων, ειδικά για τα επαπειλούμενα είδη. Τούτου λεχθέντος, οι συνάδελφοί μου είπαν κάτι που θέλω να πω κι εγώ. Ε, στην έκθεση για τη διατήρηση τη βιοπικιλότητα που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκάθαρα όχι μόνο αναγνώρισε την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απώλεια της βιοπικιλότητας, αλλά, όπως θα διαπιστώσατε, τόνισε το σημαντικό ρόλο της ε, Ευρωπαϊκή αλληλευτική πολιτική στον τομέα αυτό. Όπως ξέρετε, η θαλάσσια βιοπικιλότητα ε, πλήττεται ιδιαιτέρω. η κατάστασή τη είναι επικίνδυνη, 88% των αλλιευμάτων υπεραλλιεύονται και το 30% από αυτά βρίσκονται κάτω από τα ασφαλή όρια επιβίωσης. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να μην ξαναφτάσουν στην αρχική τους κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος για μια ολόκληρη οικονομική δραστηριότητα αλλά και για την τροφή από την οποία εξαρτώνται ολόκληροι πληθυσμοί στον πλανήτη μας. Η ευθύνη υπάρχει, το έχετε αναγνωρίσει και η πολιτική μας είναι σημαντική για το μέλλον. Κυρία Δαμανάκη, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι έχει την υποστήριξή μας για τις προσπάθειές σας, ούτω ώστε η κοινή αγγλευτική πολιτική να επιτρέψει τη διατήρηση των ειδών, αλλά και την αξιοποίηση της ε, θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η οποία θα είναι θα μα ε, εξυπηρετήσει καλύτερα αν την προστατεύσουμε περισσότερο. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Θα μπορούσατε πιο συγκεκριμένα να μα πείτε ποιε είναι οι διασμεύσει σα. για τα κριτήρια που συνδέονται με την προστασία τη βιοπικιλότητας που θα ενσωματωθούν στη μελλοντική κοινή αλληλευτική πολιτική και ποια είναι τα μέτρα τα οποία προβλέπετε να προωθήσετε για να ανακτήσουμε την ε, θαλάσσια βιοπικιλότητα στα πλαίσια αυτής της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτική. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την Επίτροπο και να την ευχαριστήσω που ήρθε να ζητήσει την υποστήριξή μας στις μελλοντικέ προσπάθειες υπέρ μιας βιώσιμης πολιτικής αλληλείας. Όταν συναντώ κόσμο και συζητώ θέματα ευρωπαϊκά, πολλές φορές παραπονιούνται διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει όλο να πηγαίνει στο Στρασβούργο και θεωρούν ότι αυτό ε, είναι ε, πολύ δυσάρεστο για την Ευρώπη. Και πάντα απαντάω και λέω δεν είδατε τι σε τι κατάσταση είναι όμως η ευρωπαϊκή πολιτική αλίας. Όχι, όχι, το λέω αλήθεια, το σοβαρό λόγο. Δεν είναι δρόμος αυτός για την Ευρώπη να ακολουθήσει. Και νομίζω ότι και εσείς το ίδιο μας είπατε ουσιαστικά και ε, είπατε ότι δεν πρέπει να παραπονούμεθα μόνο για το Συμβούλιο και τη στάση του, αλλά να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τις ε, προτάσεις σας για το μέλλον της, ε, πολιτικής, της κοινής πολιτικής οπότε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα εδώ. Μια ερώτηση όμως έχω να κάνω σχετικά με το πρόβλημα από πάνω προς τα κάτω που βλέπετε, που εντοπίζετε και ότι ε, πρέπει να κινηθούμε προς περιφερειοποίηση μάλλον. Αν δω πώς λειτουργεί τώρα η κοινή αλληλευτική πολιτική, όπου τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση, εφαρμογή και ακούω ιστορίες ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πολύ αυστηρά και δεν παίρνουν πολύ στα σοβαρά την ε, εφαρμογή. Τι θα γίνει όταν η περιφερειοποίηση ενταθεί βλέπω προβλήματα εκεί. Επίσης, δύο ακόμα για τον κοκκινό τόνο. Ήμουν στην ε, διάσκεψη ε, της Ντόχα ε, στις αρχές του χρόνου, της ΣΥΤΕΣ, και είδα ότι η Ευρώπη κάπου κατέληξε, αλλά μπλοκάρισε το δρόμο η Ιαπωνία, η οποία είπε στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν είναι οι ΣΥΤΕΣ που πρέπει να ασχοληθούν με τον κόκκινο τόνο, αλλά το ICAD, εσείς τώρα θα συμφωνήσετε ή πιστεύετε ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει με, με, με μηδενική ποσόστοση στο ICON, σε αυτό το είδος, ή θα, στην ε, ε, Μεσόγειο τι θα γίνει με τον κόκκινο τόνο, ιδιαίτερα ε, στην εποχή του. Και το σύστημα αποπληρωμών που χρησιμοποιηθεί, ότι αν ξεπεράσετε ε, μέσα σε ένα χρόνο την ποσόστοση, τότε μειώνει την ποσόστοση τον επόμενο. Το 2007 όταν μειώθηκαν οι ποσοστώσεις, η ICAT συμφώνησε για δύο χρόνια να βάλει το σύστημα ε, ε, επιστροφής στο ψυγείο, να το παγώσει και να μην το συζητήσει άλλο το θέμα της μείωσης των ποσοστώσεων. Νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί τον Νοέμβριο στη συνάντηση ICAT. Ελπίζω να με διαβεβαιώσετε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να απαντήσετε τώρα. Να ευχαριστήσω όλους σας. Οι παρεμβάσεις σας ήταν σαφείς, ολοκληρωμένες. Καταρχήν να υπογραμμίσω ότι και εγώ έχω μεγάλες προσδοκίες από τις προσπάθειες που κάνουμε για τη μεταρρύθμιση αυτή όχι επειδή εγώ η ίδια είμαι φιλόδοξη ή επειδή ξέρω καλύτερα τα πράγματα από εσά ή από οποιονδήποτε άλλον, αλλά επειδή τώρα είναι η ώρα. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, τότε το μέλλον δεν θα είναι καλό για την Ελία. Γι' αυτό ήθελα να υπάρξουν κάποιες ε, επίσημες αξιολογήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση και ζητήσαμε μία επίσημη μελέτη και αξιολόγηση επιπτώσεων της τωρινής μας πολιτικής. Πήραμε τα αποτελέσματα, δεν τα έχουμε όλα για το μέλλον, δηλαδή τι δείχνουν οι τάσεις, αλλά έχουμε ε, αποτελέσματα για την τωρινή μας πολιτική. Πήγα λοιπόν στο Συμβούλιο, πήγα και στην Κομισιόν, γιατί κάποιος ρώτησε, έθεσε το θέμα της πολιτικής στήριξης εδώ. Πήγα στην Κομισιόν λοιπόν με τα στοιχεία αυτά αυτές τις αξιολογήσεις τη επιπτώσεων, τη μελέτη επιπτώσεων. Τα στοιχεία λένε ότι αν συνεχίσουμε την υφιστάμενη πολιτική σε 10 χρόνια, το 2012 δηλαδή, μόνο 6 με 8 από τα 136 αποθέματα θα υφίστανται. Αυτή είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων δεν είναι από την Κομισιόν, με λέτε, δηλαδή δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση ή η Επιτροπή Περιβάλλοντο που τα λέει αυτά, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια επίσημη αξιολόγηση επιπτώσεων από την Κομισιόν. Οπότε το Σώμα των Επιτρόπων το συζήτησε το θέμα κάπω και αποφάσισαν οι άλλοι οι συνάδελφοι οι επίτροποι να με στηρίξουν ε, να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να το κάνουμε αυτό. Όμω, και θέλω να είμαι ειλικρινέστατη εδώ, η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει μία πρόταση. Αυτό που μπορώ να πω ε, ειλικρινά είναι ότι η πρόταση θα είναι φιλόδοξη. Βέβαια, η πρότασή μου θα υποβληθεί σε εσά και στο Συμβούλιο, και στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρότασή μου θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο, την Ολομέλεια, προφανώς όχι μόνο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα συζητηθεί με όλα τα μέλη. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη πολλών μελών αλλά, ή όλων των μελών. Αλλά έχει λόγο σοβαρό η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε αυτό το θέμα και αυτό ζητώ την υποστήριξή σας. Η πρόταση θα είναι φιλόδοξη λοιπόν. Δεν θα είναι, πώς να σας το πω, δεν θα είναι, δηλαδή θα περιοριστούμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή όλων των προτάσεων που ε, θα έχω λάβει, αλλά μετά πρέπει να πάω και στο Συμβούλιο, όπου θα χρειαστεί να διαπραγματευτώ Προφανές είναι αυτό και πρέπει να πω, επειδή έγινε και άλλη μια ερώτηση σχετικά με την κατάσταση στο Συμβούλιο, για να είμαι ειλικρινής δεν νομίζω ότι έχω και πολλούς συμμάχους εκεί. Δεν έχουμε πολλούς συμμάχους σε σχέση με υπέρ δηλαδή της επιλογής της αηφορίας και βιωσιμότητας. Αναφέρομαι στις κυβερνήσεις. Και το πρόβλημα είναι ότι ως επιτοπλίστων οι κυβερνήσεις εκπροσωπούνται από τους Υπουργούς Αλίας Καμιά φορά οι Υπουργοί Αλίας, και αυτό θέλω να σας το πω, να σας το εξομολογηθώ δηλαδή, έχω περιπτώσεις κρατών μελών όπου ο Υπουργός Αλίας είναι και Υπουργός Περιβάλλοντος. Και ακόμα και τότε οι Υπουργοί δεν τάσσονται υπέρ μιας γνήσιας περιβαλλοντικής αλλαγής. Όταν όμως είναι μόνο η Υπουργή Αλίας εκεί, τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε γιατί θέλουν να προασπίσουν ο καθένας τα συμφέροντά του. Δεν κατηγορώ, δεν, δεν παραπονιέμαι για το Συμβούλιο. Ούτε θέλω όλο το φταίξιμο να το ρίξω στο Συμβούλιο. Αυτό που είπα και θέλω να επαναλάβω είναι ότι πρόκειται για μια κοινή προσέγγιση, κοινή θεσμική προσέγγιση. Και η προσέγγιση είναι ότι πρέπει να δώσουμε λεφτά, να έχουμε μεγάλα σκάφη, να αυξάνουμε τις αλληλευτικές δυνατότητες και μετά θα πρέπει να ξαναπληρώσουμε για να ξαναρίχνονται τα ψάρια στη θάλασσα. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Έτσι σας το λέω ειλικρινά. Τι να περιμένω από το Συμβούλιο. Περιμένω από το Συμβούλιο να, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και θέλω να είμαι και εδώ πολύ ειλικρινής θα πάω με κάποιες προτάσεις για τις ποσοστώσεις του επομένου έτους και θέλω να ε, μείνω στις, ε, στα επιστημονικά δεδομένα. Το έχω πει 100 φορές και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και δεν το πιστεύουν. Κανείς δεν πιστεύει τα στοιχεία, ούτε τώρα ακόμα, 20 μέρες πριν από το Συμβούλιο. Δεν τα πιστεύουν, νομίζουν ότι μετά θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση, δώσ' μου 100 τόνους ε, μπακαλιάρου, να σου δώσω εγώ ε, ε, ρέγγα, αλλά έτσι πια δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και εδώ χρειάζομαι την υποστήριξή σας. Εγώ προτίθεμαι να πάω το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, τότε που θα πρέπει να αποφασίσουμε για τις ποσοστώσεις του χρόνου και να δώσω ένα πρώτο, να στείλω ένα πρώτο μήνυμα. Θα του πω, αυτά είναι τα περιθώρια που μου δίνει η Επιστημονική Επιτροπή. Μπορώ να επιδείξω ευελιξία και να πάω, να εξαντλήσω τα περιθώρια και να συμφωνήσουμε κάπου εκεί, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε πλέον τα επιστημονικά πορίσματα. Αν τα πορίσματα, γιατί αυτό συνέβη στο παρελθόν. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα, συγκεκριμένα παραδείγματα, αν έχω χρόνο. Για κάποια είδη, όπου για παράδειγμα μιλούσαν για 10.000 τόνους, τα επιστημονικά δεδομένα και εμείς ανεβήκαμε στους 20.000 τόνους. Και έχω υπουργού που είπαν, που λένε τάσσονται υπέρ του περιβάλλοντος και τους αρέσουν πολύ, ε, ε τους αρέσει η βιώσιμη ελία και μετά πιέζουν για αύξηση του, των τόνων. Βέβαια, ε, ε μου και καθήκον μου είναι να αντισταθώ εγώ, κανείς άλλος ε, δεν μπορεί να το κάνει ούτε λέω ότι φταίει κάποιος άλλος. Αλλά εδώ χρειάζομαι υποστήριξη για να... Γιατί το Συμβούλιο, σας το λέω, δεν αρέσκεται στις ριζικές αλλαγές. Δεν τους κατηγορώ. Έτσι δουλεύαμε μέχρι τώρα, επί σειρά ετών. Και πρέπει επίσης ειλικρινέστατα να πω ότι αντελήφθην ότι δυο φορές η Κομισιόν προσπάθησε να περάσει τη μεταρρύθμιση ε, δεν είμαι εγώ δηλαδή που είχα αυτή τη φαϊνή ιδέα, δυο πρώτη, δυο φορές επιχείρησε να κάνει μεταρρύθμιση κομισιών και απέτυχε. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Ναι στη διαπραγμάτευση, αλλά να μπορούμε να κοιταζόμαστε και να έχουμε την ε, συνείδησή μας καθαρή. Τώρα για τον κόκκινο τόνο. Ήταν πάρα πολύ απογοητευτικά και τα αποτελέσματα και οι προσπάθειες που έγιναν, το όλο εγχείρημα. Ήρθε η Ιαπωνία και μας είπε σε όλους, σε όλο τον κόσμο, ότι εμείς έχουμε την δύναμη, έχουμε και τα χρήματα. Αυτό έχουμε τώρα, αυτό, τι, μόνο το ICAD μένει ως λύση μέχρι την επόμενη συνάντηση σάιτες. Ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε είναι να πείσουμε όλους στο ICAT, να τους πείσουμε. Θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε, να παρακολουθούμε και να σεβόμεθα τα επιστημονικά δεδομένα. Τώρα, για συγκεκριμένες ποσοστώσεις δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν έχω επιστημονικά στοιχεία. Θα τα πάρω αυτή τη βδομάδα και την επόμενη βδομάδα τα περιμένω. Μόλις τα λάβω θα πω ότι στην ΆΙΚΑΤ θα ε, σεβαστούμε τα επιστημονικά πορίσματα. Αν τα επιστημονικά πορίσματα λένε να μειώσουμε την ποσόστοση, θα το κάνουμε. Και να κλείσει, ε, θα πατήσει η αλία, αν δεν υπάρχει συμμόρφωση εδώ. Επίσης, ε, τα, ε, τα ε, απειλούμενα από εξαφάνιση ήδη, ποια είναι, πώς θα αντιμετωπιστούν, σε, με προγράμματα μακράς πνοής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να δουλεύουμε μακροπρόθεσμα. Μόνο έτσι μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μαζί μας γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια θνησιμότητα ή μέγιστη ε, βιώσιμη απόδοση, ε, το προτιμώ, και μετά να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο ώστε να κάνουν και εκείνοι τις προσπάθειες που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος. Δεν είναι εύκολο αυτό. Τώρα για τον κόκκινο τόνο, το Νοέμβριο όπως είπατε, το Συμβούλιο στη, για το ICAD στο Παρίσι θα συνεδριάσει, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Οπότε εκεί θα δούμε το, αυτό το σύστημα επιστροφής ή ή σημείωσης. Ε, δεν μου αρέσει, αλλά πρέπει να ε, είμαστε συνεπείς με τις αποφάσεις μας. Πρέπει να το πω αυτό. Και να πω επίσης ότι πάμε εκεί με φιλόδοξη πρόταση ως Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να πείσουμε και του άλλους. Και κάτι άλλο που θέλω να πω σε αυτά τα πλαίσια. Μιλάμε για τον κόκκινο τόνο, υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσπάθειες ε, ε, να διατηρηθεί υγιές το απόθεμα αυτό, αλλά λέμε λίγα για τις άλλες μεσογειακές χώρες. Η Τουρκία, η Λιβύη, η Τινησία, αλλιεύουν όλοι. Και ο μόνος τρόπος ελέγχου είναι να με την ICAD να ελέγχει την κατάσταση και να αναλάβει γνήσιες πρωτοβουλίες για να διαεξασφαλίσει τη συμμόρφωση. Πράγμα καθόλου εύκολο, διότι δεν είναι κράτη-μέλη. Την άλλη εβδομάδα πάω στην Τουρκία για να πείσω τις τουρκικές αρχές ότι πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας γιατί έχουμε πολλά προβλήματα εκεί. Αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι θα τους πείσω. Πάντως οφείλω να προσπαθήσω. Τώρα για το συντονισμό μας. Αυτή είναι η πρόταση μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Αυτό που μπορώ να περιμένω από εσά, πολύ συγκεκριμένη πρόταση είναι αυτή, να συνεργαστούμε για να βρούμε με το ε, τον ειδικό θαλάσσιο σχεδιασμό, να βρούμε κάποιους τομείς σε κάθε κράτος μέλος, να ορίσουμε τις περιοχές που πρέπει να προστατεύονται για λόγους βιοπικιλότητας, ε, για λόγους ε, οτοκίας κλπ. Αυτό είναι ένα μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα βοηθηθεί πολύ η αλληλεία. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα ειλικρινά να ελέγχουμε επακριβώς το σύστημα των ποσοστώσεων. Γιατί έχουμε τις εκφορτώσεις, τις απορρίψεις, τα λιεύματα, είναι περίπλοκο. Αν κλείσουμε όμως μια περιοχή για λόγους οτοκίας, αναπαραγωγής, για μια-δυο σεζόν, τότε μπορούμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα εκεί, γιατί εύκολα ελέγχεται η περιοχή. Η κλειστή περιοχή είναι πιο εύκολο να ελέγχεται, με πάση περιπτώσει, δεν θα πάει κανείς να ψαρεύει εκεί. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε εκεί και να πείσουμε τις κυβερνήσεις να το κάνουν. Μέσα από την οδηγία για τις θαλάσσιες, θαλάσσιες υποθέσεις να ορίσουν τις περιοχές, να τις κλείσουν και να θεσπίσουν κανόνες προστασίας τους. Τώρα για την περιφερειοποίηση και τη συμμόρφωση, αυτό αφορά μια άλλη ερώτηση, Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη συμμόρφωση, γιατί η πολιτική είναι πολύ σύνθετη και πολύπλοκη. Μια απλούστερη πολιτική θα δίνει καλύτερη, καλύτερο ποσοστό εφαρμογής. Έχουμε όμως νέα όπλα με τον κανονισμό τον καινούριο, τον Αγίου. Μπορούμε να ε, προσφύγομαι κατά των κρατών μελών. Από την 1η Ιανουαρίου έχω καινούριο όπλο κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Και θα το εφαρμόσω. Επίσης, η περιφερειοποίηση στόχο έχει να αυξήσει την υπευθυνότητα του τομέα και της, των περιφερειών μας. Και ξέρω πολύ καλά ότι οι περιφέρειες μπορούν να οργανώσουν τη συμμόρφωση καλύτερα, γιατί γνωρίζουν τι συμβαίνει στην περιοχή τους σε μικρότερη περιοχή οι αρχές γνωρίζουν καλύτερα τι συμβαίνει και μπορούν, εφόσον έχουν τη βούληση, προϋπόθεση είναι αυτό, μπορούν να διασφαλίσουν την συμμόρφωση που θέλουμε. Έτσι βλέπουμε εμείς την περιφερειοποίηση. Και τέλος, για τις ε, συμφωνίες, τις ελευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, αυτό είναι ένα κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής, Είπα ότι πρέπει να ε, διευρύνουμε τις, ε, και, να, και να μεταλαμπαδεύσουμε δηλαδή τις αρχές μας παντού, γιατί είμαστε εισαγωγή πολύ μεγάλη, πρέπει να πείσουμε τις χώρες που εξάγουν ε, ψάρια ότι πρέπει να δουλεύουμε με βιώσιμο αηφόρο τρόπο και θα πρέπει αυτό να ισχύει γενικότερα στις εισαγωγές. Και πρέπει να ισχύει και στι αγωγέ, δηλαδή το νέο σύστημα, όχι μόνο στα δικά μα αλλιεύματα. Ελπίζω να μπορέσω να πείσω τους ε, συναδέλφους μου επιτρόπους να έχουμε μια κοινή πρωτοβουλία εδώ. Και περνώ στι αλλιευτικέ συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Θέλουμε για το αλλιεία του πλεονάσματο στι περιοχές που πηγαίνουμε. Πρέπει να πω ότι ε, δεν ισχύει αυτό πάντοτε και πολλές φορές έχουμε προβλήματα με τον τόπιο πληθυσμό. Η, μία από τις, η δεύτερη σε σημασία τέτοια συμφωνία είναι με το Μαρόκο. Και αυτή συνοδεύεται από ένα πρωτόκολλο που λύγει τέλος Ιανουαρίου, εκπνέει η συμφωνία, το πρωτόκολλο και μέχρι τώρα δεν έχω αναλάβει πρωτοβουλία ανανέωσης γιατί η μαροκινή κυβέρνηση δεν είναι συνεργάσιμη και δεν μας δίνει όλα τα στοιχεία για τους ε, δικαιούχους, τους ντόπιου πληθυσμούς στο δυτικό Μαρόκο δεν μας δίνει στοιχεία για τον πληθυσμό εκεί. Θέλουμε να επιληθεί με το σωστό τρόπο το πρόβλημα. Τους έδωσα μια τελευταία διορία να μας τα στείλουν και θα υποβάλω την πρότασή μου, συγκεκριμένες δηλαδή προτάσεις, στην Επιτροπή Αλίας μετά από δύο εβδομάδες τότε θα είμαι έτοιμη να υποβάλω συγκεκριμένη πρόταση για τη συμφωνία αυτή και το πρωτόκολλό της. Γιατί με, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ευτυχείς από τη συμφωνία αυτή. Το λέω για να σας, το, αυτό για να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Χρειάζεται αλλαγή εδώ και πρόθεσή μου είναι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ε, πολιτικής ελίας να έχουμε νέο κεφάλαιο για την εξωτερική πολιτική και τη Συμφωνία Ελίας, ένα κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες με τις οποίες ε, συναλλασσόμεθα και πάμε και αλλιεύουμε εκεί και θέλουμε και καλή συμμόρφωση για ε, τον κόσμο εκεί και τους πραγματικούς δικαιούχους των χρημάτων που δίνουμε, γιατί τα ποσά είναι μεγάλα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλού τομεί. Ε, η πολιτική αυτή είναι μικρή, λέει η κυρία Δαμανάκη, παρόλα αυτά έχει πολλέ πτυχέ. Υπάρχουν ε, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πτυχές αυτής της πολιτικής με μεγάλο ενδιαφέρον σας ακούσαμε. Έχουμε και άλλους ομιλητές, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο κύριος Πανιό. Δύο-τρία λεπτά ο καθένας σας παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ναι, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση για το Μαρόκο ακριβώς. Μόλις ε, μιλήσατε για το θέμα αυτό του Μαρόκου, για την ανανέωση της ε, αληφτικής συμφωνίας με το Μαρόκο, η οποία εκπνέει τον ε, Ιανουάριο του 2011, όπως είπατε. Στα πλαίσια μια συνεδρίαση που έγινε τον Ιούλιο φέτος, είπατε εσείς ότι σκοπεύατε να πάρετε την απόφαση τέλος Αυγούστου. Τώρα έχουμε φτάσει τέλος Σεπτεμβρίου. Θα σας πρότεινα λοιπόν να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα, πού έχετε φτάσει. Είναι 27-28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τι αποφάσεις έχετε πάρει, σας παρα... πέστε μας σας παρακαλώ. Επίσης, θα έρθω σε επαφή με τον, ε, αυτό το Σάββατο με τον Υπουργό ε, Αλίας του Μαρόκου για να συζητήσω και πολιτικά θέματα και προσωπικά θέματα βέβαια και αν θέλετε δεδομένης αυτής τη συνάντηση που θα έχω το ε, Σάββατο το μεσημέρι μαζί του μήπως θα μπορούσα να σας βοηθήσω ίσως ούτως ώστε να του περάσω ένα μήνυμα ιδιαίτερο ούτως ώστε να σας ενημερώσω μετά για τις απαντήσεις του. Μια και μας είπατε ότι θα πάρετε προσεχώς μια απόφαση τις επόμενες 15 μέρες. Να μια προσφορά. Υπάρχουν και, άλλες, υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερες σχέσεις με το Μαρόκο. Μπορεί να σας βοηθήσει αυτό. Μοκονάιτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Το ερώτημά μου αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση να αυξήσει τις ποσοστώσεις του γάδου που ψαρεύεται στη Βαλτική. Η απόφαση βασίστηκε υποτίθεται σε επιστημονικά δεδομένα. Αλλά όμως η Βαλτική θάλασσα είναι πολύ μολυσμένη. Το πλανκτόν είναι στα όρια Τη ακύρωση. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Επομένως, τι θα φάνε τα ψάρια. Και το, τα ψάρια αδυνατίζουν και γίνονται όλο και λιγότερα. Υπερβαίνουμε μάλιστα τις ποσοστώσεις κατά πολύ. Κατά πολύ. Όταν λοιπόν λήφθη αυτή η απόφαση, λάβατε, λάβατε υπόψη αυτήν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι είδατε τα επιστημονικά στοιχεία. Ε, όταν μιλάμε για τη μόλυνση, τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν και αυτά την προετοιμασία τους, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει σχετικές προτάσεις. Καλή είναι η μεταρρύθμιση των πολιτικών, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα νερά μας είναι πολύ μολυσμένα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι που ακούγονται και ανησυχίες που ακούγονται για την ποιότητα των ψαριών μας. Η Φρανσουάς Γκοστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, μας είπατε πολλά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να επανέλθω στο εξή. Έχουμε μια υπεραλίευση. Κανένα δεν σέβεται ουσιαστικά τι ποσοστώσει σήμερα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές ενισχύσει επίσης που δίδονται για να υποστηρίξουμε όχι μόνο το βιώσιμο, μια, ένα βιώσιμο αλληλευτικό στόλο, αλλά έναν αλληλευτικό στόλο που δεν σέβεται τελικά τις δεσμεύσεις μας για το περιβάλλον. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι δεδομένα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δυσκολίες. Θέλουμε υποτίθεται να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα και τα είδη. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ε, θέσεις απασχόλησης επίσης που εξαφανίστηκαν και άλλες που απειλούνται. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Σας ευχηστώ την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την παράκτη αλία. Το είπατε. Είπατε ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτή την αλία, αυτή που συμμετέχει στην οικονομική ζωή των ακτών μας και που είναι πάρα πολύ σημαντική αλληλεία. Έχουμε εδώ και δεκαετίες, μια και υπάρχει φοβερή ανισορροπία μεταξύ της παράκτιας αλληλείας ή όπως λέγεται εραστεχνικής και της βιομηχανικής ή εκτατικής, ε, εντατικής, συχνά θυσιάζουμε αυτούς τους μικρούς αλληλείς στο βωμό της βιομηχανικής μεγάλης έκτασης αλληλεία. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και αβιώσιμη ανάπτυξη, μην ξεχνάμε αυτού του ανθρώπου, αυτού του αλλεί, αυτή την αλία. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να υποστηρίξετε αυτή την παράκτη αλία. Και επίση, τι ρόλο θα έχει η χθιοκαλλιέργεια. Επί μακρόν λέγαμε ότι η χθιοκαλλιέργεια θα μπορούσε να είναι πανάκια για να αντικαταστήσει μάλιστα και να υποκαταστήσει κάποιου είδου αλία, ειδικά στα ευαίσθητα είδη, στα ευάλωτα είδη. Αλλά και εκεί υπάρχουν παραβιάσεις, παραβάσεις, προβλήματα, ε, δημιουργούνται υγειονομικά προβλήματα και προβλήματα διαχείρισης της ηχθειοκαλλιέργειας. Τι πιστεύετε για την περιβαλλοντική επίπτωση της ηχθειοκαλλιέργειας. Βαραίνει το περιβάλλον. Ποια είναι η άποψή σας. Επίσης μιλήσαμε για τις ε, αληφτικέ συμφωνίες με τρίτες χώρες. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν θα θυσιάζουμε τους δικούς μας αλληλείς και θα ευνοούμε τους ξένους. Ευχαριστώ τη Φρανσουά Γκροστέτ. Μαρίτα ε, Ευχαριστώ για την παρουσία σας, κυρία Επίτροπε. Το θέμα της αλίας απασχολεί και τη δική μας Επιτροπή. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Άκουσα τις παρουσιάσεις σας. Άκουσα την, αυτό που είπατε για την αντίδραση των ενδιαφερομένων φορέων και για την αντίδραση των Υπουργών Αλίας, οι οποίοι αγνοούν τις καταστροφές που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πρόκειται περί καταστροφών. Υπάρχουν επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στο κλίμα. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα ανοιχτά. και όμως τόσοι πολιτικοί κλείνουν τα μάτια μπροστά σε αυτή την καταστροφή, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Αγνοούν και κλείνουν τα μάτια μπροστά στα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε επιτάπητος. Αγνοούν τις προκλήσεις, παρότι η καταστροφή είναι πρώτων πυλών. Ορισμένοι ακόμα εθελοτυφλούν. Άκουσα τις ερωτήσεις, άκουσα και τις απαντήσεις που δώσατε και με μεγάλη χαρά σας, σας άκουσα να λέτε ότι θέλετε να προωθήσετε μία συνολική μεταρρύθμιση. Μία πλατιά και βαθιά μεταρρύθμιση. Η Βαλτική δεν είναι τόσο μεγάλη θάλασσα σε σχέση με άλλες θάλασσες στην, στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συνάδελφος αναφέρθηκε στην καταστροφή που λαμβάνει η χώρα στη Βαλτική, στο εσωτερικό αυτής της θάλασσας. Είναι μια θάλασσα ε, η οποία είναι αρκετά κλειστή. Δεν μπαίνω βγαίνει πολύ νερό. Επίσης είναι και η φάλμηρη η θάλασσα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους αλείς οι οποίοι παρέλαβαν τη σκητάλη από τους ε, προγόνους τους, από τους πατέρες και παππούδες τους. Κι όμως σήμερα υπάρχουν πολλοί που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Χρειαζόμαστε λιγότερα βέβαια αλληλευτικά σκάφη και λιγότερους ανθρώπους που αλλιεύουν. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι το εξή. Τι δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, θα, οι οποίοι θα πρέπει να οδηγηθούν προ άλλου ε, οικονομικούς τομεί, προ άλλη δραστηριότητα αν θέλουν να παραμείνουν σε αυτές τις παράκτιες περιοχές. Εκεί σε αυτές τις ίδιες περιοχές μπορούν να δουλέψουν αλλού. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μην μετακινηθούν από τις περιοχές τους τουλάχιστον, παρότι θα αλλάξουν επάγγελμα. Ελτζαπέντα Τζαρντίνη, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή, είμαι Ιταλίδα και το πρόβλημα αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί έχουμε χιλιόμετρα ακτών και πολλές ε, περιοχές γύρω από τη θάλασσα που ασχολούνται από αρχαιοτά τον χρόνο με αυτή τη δραστηριότητα. Όταν μιλάμε για τον ερυθρό τόνο, έχετε κάποιες ιδιαίτερες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύεται εδώ και αιώνες ο ερυθρός τόνος. Υπάρχουν ε, επιστημονικά στοιχεία για μη ε, διεισδυτικέ τεχνικές που είναι συμβατές με τα οικοσυστήματα και που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Για τον ερυθρό τόνο μιλάω. Επίσης, μπορούμε τα τάκ να τα συνδυάσουμε με πιο οικολογικές προσεγγίσεις. Είπατε ότι αυτή η προσέγγιση που έχουμε από πάνω προς τα κάτω συχνά είναι η αιτία της διαιώνισης των προβλημάτων μας. Γιατί είναι ακατάλληλος τρόπος για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Θέλω λοιπόν να καταλάβω αν υπάρχουν σχέδια ανάκτησης, ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση σε κάποια είδη τα οποία έχουν υπεραλειφθεί. κάποιες περαιτέρω εξηγήσει για το πρόβλημα των ληφτικών στόλων. Σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, τα μέτρα που ρυθμίζουν τις δημόσιες ενισχύσει για την κατάργηση και καταστροφή των σκαφών δεν διαφοροποιούν ανάμεσα στα διαφορετικά σκάφη. Δηλαδή ανάμεσα στα μικρά, ας πούμε, όπου στην Ιταλία, Φερρυπίν, είναι πάνω από το 80% των συνολικών σκαφών από τη μία λοιπόν και από την άλλη τα μεγάλα σκάφη, τα βιομηχανικά αν θέλετε, τα οποία είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στις κοινότητες των αλλιέων, οικονομικά και άλλα. Για όλους αυτούς τους λόγους άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόθεσή σας για την αναδιοργάνωση της ΚΟΑ. Μιλήσατε για κάτι πολύ σημαντικό, την ετικετοθεσία επίσης, την επισήμανση. Επίσης θα δώσετε σημασία στην ε, τιμή, την πρώτη τιμή, της πρώτης πώληση, καθώς και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ε, οι οποίες ε, εισαγωγές στάνουν με ελάχιστους δασμούς που πραγματικά ανταγωνίζονται και καταστρέφουν, ας πούμε, τη δική μας παραγωγή. Επίσης, κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τη μελλοντική χρηματοδότηση. Είπατε ότι θα υπάρξουν κανόνες Ούτω ή άλλω, ε, από την 1η Ιανουαρίου ε, υπάρχει κανόνα ότι δεν θα χρηματοδοτούμε χώρε που δεν σέβονται του κανόνε. Αν ξέρετε Μπορείτε να μας πείτε ε, σε ποιο βαθμό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε οικονομικά ενώ την αλία. Ευχαριστώ. Σα του χάσει. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο που ήρθε στην Επιτροπή μας για να συζητήσει μαζί μας τα θέματα αυτά και για την πολύ ξεκάθαρη τοποθέτησή της. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για την ε, υπεραλίευση, αυτό που έθεσε η κυρία είτε για την Βαλτική. Συνήθω μιλάμε είτε για τη Μεσόγειο είτε για τον Ατλαντικό όταν συζητάμε για υπεραλίευση. Η υπεραλίευση όμω στη Βαλτική θέτει ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, σχετίζεται με ειδικά ζητήματα. Όταν έχουμε υπεραλίευση σολομού, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται το εισόδημα και οι δυνατότητες ε, εργασίας για τις τοπικές κοινότητες ε, που ζουν ε, στον ποταμό γύρω κοντά εκεί που κινούνται αυτά τα ψάρια. Και έχω λάβει πάρα πολλά email από άτομα που ζουν γύρω στον ποταμό Τόρνιο Νιοκή, που είναι ο μεγαλύτερος ε, από τους μεγαλύτερους ποταμούς. Δυστυχώς όμως ε, εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα με την αλίευση του Σολομού. Και υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Έχει υπολογιστεί ότι η οικονομική αξία για την κοινωνία γενικότερα για τα ψάρια τα οποία πηγαίνουν στον ποταμό είναι εκατονταπλάσια τουλάχιστον σε σχέση με τα ψάρια που αλλιεύονται στη θάλασσα. Και ένα άλλο πρόβλημα σχετίζεται με την ε, υπεραλίευση που σχετίζεται με την υπεραλίευση στη Βαλτική είναι ευτροφισμός. Η Βαλτική είναι μία από τις ε, πιο μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο. Και αυτό οφείλεται στον ευτροφισμό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν ε, πρακτικά αλλιευτικά είδη τα οποία προκαλούν αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά. Δεν υπάρχουν όμως αρκετά μεγάλα αρπακτικά, παραδείγματο χάρη, τα οποία θα τρώνε ψάρια όπως η ρέγγα, που αυτό το είδος ε, ουσιαστικά έχει αυξηθεί σημαντικά, καταναλώνει το πλανκτόν, που το ε, πλανκτόν μειώνεται και έχουμε πραγματική ε, έκρηξη των τοξικών φυκιών των αλγών στην επιφάνεια της θάλασσας, αυτό το πράσινο που βλέπουμε πάνω στο νερό, στην επιφάνεια. Τι σκέφτεστε για να αντιμετωπίσετε αυτά τα ειδικά προβλήματα με την αλία στη Βαλτική θάλασσα. Merci. Julie Gelling. Ευχαριστώ, Julie Gelling. Thank you, Chairman. Um... Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, στην εισαγωγή σας Μιλήσατε για την παρακολούθηση της μικρής κλίμακας αλίας, ότι θα ελέγξετε από κοντά την κατάσταση. Θα ήθελα να μας πείτε πώς προχωρεί αυτή η έρευνα, ποιες προοπτικές βλέπετε να υπάρχουν για την υιοθέτηση ενός διαφοροποιημένου καθεστώτος για τον στόλο αυτό, τον αλλιευτικό, γιατί πραγματικά σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή παράκτη αλία που ανέφεραν και άλλοι, είναι κάτι πολύ σημαντικό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μια άλλη ερώτηση. Δεν μπορώ ε, να εκπροσωπήσω τους Βρετανούς αλληλείς αν δεν αναφέρω ε, το ζήτημα που έχουμε με τις νήσους ε, Φερόε σε σχέση με τον Βακαλάο. Και έτσι μπαίνει στο επίκεντρο, μπαίνει στο προσκήνιο το πρόβλημα με τις συμφωνίες τις εξωτερικές και την εξέβρεση εταίρων και με την κυβέρνηση των Ίσων Φερό αλλά και με την Ισλανδική κυβέρνηση έχουμε προβλήματα, δεν μειώνουν τα λεύματά τους, είναι πάρα πολύ υψηλά, ε, αστρονομικά υψηλά θα έλεγα και θα ήθελα να μας πείτε αν στη νέα πολιτική την οποία εκπονείτε θα υπάρχουν πάρα πολύ πιο αυστηροί κανόνες, θα υπάρχουν τρόποι για την εφαρμογή, για την επιβολή των κανόνων αυτών. Ο κύριος Κυλακάκης έχει Κυρία Επιτρόπε, ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική ε, παρουσίαση. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο είναι το θέμα της παράκτειας σε σχέση με την βιομηχανική αλία. Το έθεσε και η Σάτου Χάση. Ε, αναφερόμενοι στους ποταμούς, εγώ θα το θέσω αναφερόμενη στις τουριστικές, αναφερόμενος στις τουριστικές περιοχές. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι τα ε, ψάρια που ψαρεύονται από την παράκτη αλία σε, ε, σε τουριστικές περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Και πρέπει να βρούμε τρόπους για να προστατεύσουμε την παράκτη αλία από την βιομηχανική αλία. Ε, διότι τα, τα ψάρια δεν είναι ε, ένας πόρος σε αυθονία. Δεν υπάρχουν άλλωστε πια στον πλανήτη πόροι σε αυθονία, ούτε ο αέρας όπως έχουμε ανακαλύψει δεν είναι σε αυθονία πόρος. Είναι ένας πεπερασμένος πόρος και κάποιος ο οποίος υπεραλλιεύει το κάνει αυτό εις βάρος του συνολικού κοινωνικού συνόλου. Το δεύτερο θέμα που ήθελα να θέσω αφορά τις ηχθειοκαλλιέργειες και έναν φόβο ο οποίος υπάρχει και θα ήθελα να σας προβληματίσει για την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών στις ηχθειοκαλλιέργειες. Η ε, υπερβολική χρήση αντιβιωτικών κρύβει πολύ μεγάλους κινδύνους γενικότερα. Ε, το έχουμε αυτό ε, στα νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς εκτός της ανθρώπινης υγείας, όπου χρησιμοποιούνται μαζικά αντιβιωτικά και στην περίπτωση των ηχθειοκαλλιεργιών, επειδή είναι δύσκολο να δώσει στα ψάρια αντιβιωτικά ένα-ένα, μιλάμε για μαζική χρήση. Και το τρίτο θέμα που ήθελα να θέσω ε, αφορά ε, την, τάση για στροφή στην περιφερειακή, ε, αν θέλετε, οργάνωση της, των του, ελέγχου και της επιβολής ε, του compliance, της επιβολής της νομοθεσίας. Ε, έχω αμφιβολίες για το αν μια μαζική στροφή προς την περιφέρεια είναι ό,τι καλύτερο. Και αμφιβολίες μου δράζονται στο εξής. Το πολιτικό σύστημα το περιφερειακό έχει πολύ μεγαλύτερες επιρροές των αυτών που ψαρεύουν και πολύ μικρότερες επιρροές των, ε, αυτών που αναφέρονται για το περιβάλλον. Διότι καλός ή κακός σε όλη την Ευρώπη, στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει πολύ ισχυρότερη, ε, ισχυρότερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Οπότε θα ήθελα να σας προβληματίσει αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λέει ο κύριος Ρώση, το θέμα δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τη μείωση των ποσοστώσεων και τη μείωση των ζωνών και να μην μιλάμε καθόλου για την προστασία αυτής της δραστηριότητας και ότι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα γιατί θα υποστούν ζημίες. Εγώ έχω ανέβει σε σκάφος Ξέρετε πολύ καλά, ε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε ανέβει σε σκάφος, ε, ξέρετε πάντως ότι μερικές φορές ε, όταν ε, ξεφορτώνται τα δίχτυα πάνω στο σκάφος, συχνά το 90% των ψαριών πρέπει να απορριφθεί μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν είναι κατάλληλο. Παρόλα αυτά, αυτό το 90% των ψαριών που ρίχνεται μέσα στη θάλασσα είναι ήδη νεκρό. Το τα περισσότερα ψάρια είναι νεκρά. Γιατί τα έχουν, πατήσει, ε, τα έχουν πατήσει τα άλλα, γιατί είναι μικρά ας πούμε και συγκλείβονται από τα πιο μεγάλα. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να ψαρεύουμε μόνο τα μεγάλα ψάρια, αλλά ούτως ή άλλως καταστρέφονται και τα μικρά. Γιατί να μην επιμένουμε στις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και να σκεφτούμε και την Νορβηγία η οποία ψαρεύει ακόμα φάλαινες, ας πούμε. Επίσης, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ισλανδία δίνουν μάχες αλλιευτικές για τον Βακαλάου. Το είπατε κι εσείς. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε κοινούς κανόνες. Επίσης, μπορούμε να έχουμε θύλακες στο, στη θάλασσα, όπου μπορούν εκεί τα ψάρια να μπορούν να, να παράγονται. Με δίχτυα, πραγματικά προστατευμένη η περιοχή. Και από πολύ λίγα ψάρια μπορούμε να τα βοηθήσουμε να πολλαπλασιαστούν. Φυσικά κοστίζει. Αλλά κοστίζει και το να αφήνουμε ανενεργά τα σκάφη μας ίσως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για να υπάρξει αναπαραγωγή του, των ψαριών. Όχι μόνο με την καλλιέργεια, αλλά με μία ε, καλλιέργεια ψαριών στις θάλασσες, ε, αυτά τα είδη μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να, βοηθήσουμε τη θάλασσα να ξαναγεμίσει ψάρια από αυτές τις προστατευμένες ζώνες. Thank you, chairman, before you <laughs> τελευταίο ομιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε πριν φύγετε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε και μας δώσατε σαφέστατες ιδέες για την ατζέντα σας. Συγκεκριμένη ερώτηση ε, σχετικά με την ε, διάσκεψη της ΩΣΦΑ στην ε, Νορβηγία. Το ξέρετε αυτό. Τα τελευταία νέα εκεί είναι ότι υπάρχουν ε, πέντε θαλάσσιες περιοχές που έχουν οριστεί και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι τα ε, πρώτα MPAs ανοιχτή θάλασσας, οπότε αυτό είναι καλό από την ΟΣΠΑ ε, επιτέλους και επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέλος της ΟΣΠΑ, σας ερωτώ κυρία Επίτροπε, τι συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις προβλέπετε για να εφαρμοστούν τα 5 MPA όπως τα αναφέρατε και πριν. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε τις ιδέες σας σε σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής ώστε να έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα από την ε, συμφωνία αυτή, από την Ορβηγία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ότι υπάρχει εντονότατο, ζωηρότατο ενδιαφέρον, κυρία Επίτροπε. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω και να καλύψω στον δυνατόν περισσότερες πτυχές σας. Ξεκινήσω λοιπόν ε, με το Μαρόκο. Πολύ σωστές πληροφορίες που έχετε, είστε πολύ καλά ενημερωμένο. Πράγματι είχα πει τον Ιούλιο ότι χρειάζομαι κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση του Μαρόκου για τους πραγματικούς δικαιούχους της συμφωνίας μας, ιδίως ε, στο Δυτικό Μαρόκο. Περίμενα απάντηση. Λυπούμε, αλλά μέχρι στιγμής απάντηση δεν υπάρχει. Άρα ο Μαροκινός υπουργό που θα συναντήσετε δεν έχει απαντήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα του δώσω λοιπόν πώς να το πω ακριβώς, ε, θα ξαναήθω σε επαφή μαζί του και θα του πω, κοιτάξτε, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, Εξού και αναβάλω την λήψη της απόφασης. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ε, για να μην ειλικρινή σας το λέω αυτό. Και ίσως μπορούμε να έχουμε, πώς να σας το πω, να ορίσουμε μια άλλη ημερομηνία. Και αν μας ε, δώσουν πληροφορίες μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους, αλλιώς θα πρέπει να σταματήσουμε. Είναι σαφής η επιλογή, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Άρα αναβάλουμε την απόφαση μόνο και μόνο για να πείσουμε τους πάντες ε, και δει τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται για τη συμφωνία αυτή και ιδιαίτερα Γαλλία, Ισπανία και κάποια άλλα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται για τη συμφωνία αυτή με το Μαρόκο. Να πείσουμε λοιπόν αυτά τα κράτη ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για να ανανεώσουμε το πρωτόκολλο. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν μετά διαβιβάσετε το μήνυμα αυτό. Είναι σαφές. Σας στείλαμε μια επιστολή, περιμένουμε απάντηση. Εγώ ουσιαστικά ε, λέω ότι είναι θέμα όχι απλά ευγένεια για να απαντήσουν, είναι θέμα ανάγκη, είναι πήγον. Ε, είναι γραμμένο και στη συμφωνία. Δεν ζητάω πράγματα που έχω βγάλει το κεφάλι μου. Γράφεται σε συμφωνία. Προβλέπεται σε συμφωνία ότι θα πρέπει να μα δώσουν στοιχεία για του πραγματικού δικαιούχου τη συμφωνία. Αυτό ζητάμε. Και πραγματικά θα χαρώ ιδιαίτερο και αν διαβάσετε το μήνυμά μου και αν μου μεταφέρετε και κάποια είδηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι εξωτερικέ σχέσει, α ε, έλθουμε για λίγο στην Ισλανδία, στις Νουσφερόε και το θέμα του Βακαλάου. Είχαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό, μπορεί και να το γνωρίζετε. Το πρόβλημα εδώ είναι ξεκάθαρο. Με τα κράτη αυτά, Φερό και Ισλανδία, έχουμε το εξής: Έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις τους μονομερός για το βακαλά, χωρίς δηλαδή να μας ενημερώσουν, δεν μας έδωσαν καμία απολύτως πληροφορία. Τα Φερό, που είναι και μια μικρή χώρα, τριπλασίασε την ποσόστοσή τη. Καταλαβαίνετε ότι η αύξηση αυτή είναι τεράστια. Δεν μπορούμε να τη δεχθούμε. Πρέπει λοιπόν να πάμε εκεί και να διαπραγματευτούμε. Αυτό κάνουμε. Τώρα όμως έχω μια εντολή. Πήγα εκεί, συζήτησα. Τώρα λοιπόν έχω εντολή από το Συμβούλιο σε περίπτωση, ελπίζω να μην χρειαστεί, αλλά σε περίπτωση που η Σλαβία και Φερόε δεν δείξουν ευελιξία, θα πρέπει εγώ να διερευνήσω κάθε περιθώριο δράσης που έχω. Να δω όλες τις επιλογές που έχω. Ξετάσουμε λοιπόν τις ελληνικές συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με τις χώρες αυτές. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Και αυτό όχι γιατί πρόκειται για το βακαλάο, αλλά γιατί μπορεί να δημιουργηθεί προηγούμενο για εμάς με τον τρόπο αυτό. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προστατεύσει πραγματικά τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων, να προστατεύσει τη συμμόρφωση της δικής μας βιομηχανίας, του δικού μας κλάδου με τους κανόνες, πρέπει να απαιτήσουμε και από τους συμμάχους μας, από τους γειτονές μας, πείτε το όπως θέλετε, να σέβονται τους δικούς μας κανόνες. Και θα θέλαμε βέβαια να σεβαστεί η Ισλανδία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι υπάρχει τώρα ε, διαδικασία για την προσχώρηση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να συνδέσω βέβαια το θέμα της ένταξης με την αλληλευτική συμφωνία. Πρέπει να σέβονται όμως το, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για την Βαλτική έχω πάει και την έχω δει τη Βαλτική. Έχω προσωπική πείρα, έχω συζητήσει με πολλά άτομα, με αλληλείς, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ρήπανση και πολλά από τα προβλήματα τα αναφέρατε κι εσείς έχουν να κάνουν, ε, είναι μάλλον ε, αρμοδιότητα του Επιτρόπου Ποτότσνικ που δεν θέλω να υποκαταστήσω εδώ. Σε ό,τι αφορά την αλία όμως ε, θα επιμείνω στις επιστημονικές συμβουλές που λαμβάνω γιατί έτσι είμαι και αξιόπιστη. Αν εμένω και βασίζομαι στις επιστημονικές συμβουλές και υποδείξεις έχω και αξιοπιστία. Αν μας έλεγε η επιστημονική συμβουλή ότι μπορούμε να αυξήσουμε την ποσόστοση του βακαλάου, του γάδου μάλλον, στην ε, Βαλτική. Δεν μπορώ να την αγνοήσω αυτή τη συμβουλή των επιστημόνων. Μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ, ούτε θέλω να υποτιμήσω τη δική σας προσέγγιση, αλλά Υπάρχει κανόνας και πρέπει να εμείνω σε αυτόν. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα αντικρώμενα συμφέροντα στην περιοχή. Έτσι πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να ακολουθήσω την επιστημονική συμβουλή. Άλλωστε δεν πρόκειται για μια τεράστια αύξηση, νομίζω είναι τη στο του 10%. Πρέπει να γίνει όμως. Έτσι λένε οι επιστημονικές συμβουλές. Και στο κάτω-κάτω θα πάω ε, στη Βαλτική. Έχουμε τα αποθέματα ρέγκας και άλλα αποθέματα που εκεί απαιτείται μεγάλη μείωση των ποσοστώσεων για τα, για τα αποθέματα. Πρέπει λοιπόν να τους πείσω ότι πρέπει να συνεργαστούν μαζί μου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις στη Βαλτική και αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχουμε για τη Βαλτική θάλασσα. Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες ε, και τον κύριο Ποτότσιν και συγκεκριμένα, διότι πολλά από τα στήματα που αναφέρθηκαν γιατί ο ευτροφισμός και άλλα πράγματα που αναφέρατε είναι δική του αρμοδιότητας. Λυπούμε, δεν έχω στοιχεία για να σας μεταφέρω εδώ, απλά μπορώ να σας πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τις επιστημονικές συμβολές, συμβουλές ό,τι αφορά τις ποσοστός. Τώρα για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να αναδιοργανωθεί ο κλάδος. Αυτό είναι ε, η πραγματικότητα. Συμφωνώ με ορισμένους προλαλήσαντες βουλευτές για τον τρόπο με τον οποίο είχαμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε τη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, δώσαμε πολλά, πραγματικά πολλά χρήματα για την αποσυναρμολόγηση, τη διάλυση πλοίων και μετά θέλαμε να ε, ε, δώσουμε χρήματα για την ε, ναυπήγηση νέων αλλιευτικών σκαφών που δεν είχαν ψάρια να ψαρέψουν όμως αυτά τα νέα σκάφη, τα νέα πλοία. Πρέπει λοιπόν, ναι, να υπάρχει μια νέα χρηματοδότηση αλλά μόνο για μια πιο οικολογική πολιτική, μόνο για λόγους βιωσιμότητας, για την επιλογή ελευτικών ε, εργαλείων και σκαφών, για τη συμμόρφωση του ελευτικού στόλου με τους κανόνες που έχουμε. Αυτό θα κάνουμε. Πρόκειται να εγκαταλείψουμε και αυτό είναι μια απόφαση που έχει τίμημα. Σας διαβεβαιώ. Θα εγκαταλείψουμε τη χρηματοδότηση για την διάλυση σκαφών στο μέλλον. Θα εγκαταλείψουμε τη χρηματοδότηση αυτή. Υπάρχουν αντιρρήσει και αντιδράσει, αλλά δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση για άλλου σκοπού. Θα γίνει λοιπόν και η μεταρρύθμιση τη ΚΟΑ, το είπατε, αρκετοί βουλευτέ, και αυτό που χρειάζεται εδώ δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στου αλληλείς ε, για να ξαναπετάνε τα ψάρια στη θάλασσα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και εδώ έχουμε αντιδράσει πολλές αντιδράσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τα χρήματα και να βοηθήσουμε τις ε, οργανώσεις των παραγωγών, ιδιαίτερα ε, τις οργανώσεις των παραγωγών, αν είναι καλά οργανωμένοι, για να δημιουργήσουν κάποιους μηχανισμούς αποθήκευση, για να έχουν τη δική τους πολιτική αγορά και εμπορίας και να έχουν τα ψάρια, να, τα, να μπορούν να τα πουλήσουν ουσιαστικά. Δηλαδή να αλλιεύουν οι αλλοίς μας μόνο όσα ψάρια μπορούν να πουλήσουν σε καλή τιμή για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η πορεία υπάρχει. Θέλουμε λοιπόν ε, τα ψάρια που αλλιεύονται να προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Πρέπει όμως να ακολουθήσουμε μία λογική ε, αλληλουχία ενεργειών μηχανισμοί αποθήκευσης, ε, πολιτική εμπορίας ε, για να βλέπουν τι μπορούν να ψαρεύουν κτλ. Και θέλουμε να υπάρχουν ε, και ισότιμοι όροι. Θα προσπαθήσουμε, δεν είναι μου αρμόδια, θα προσπαθήσουμε πάντως να υπάρχουν ισότιμοι όροι μεταξύ των εισαγόμενων ψαριών και αυτών που ψαρεύονται στα δικά μας ύδατα να υπάρχει ένα ισοδύναμο επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά την επισήμανση, την οτικετοθεσία, επειδή είμαι βέβαιη ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής θέλει να καταναλώνει νοπό ε, ψάρι που δεν είναι ε, κατεψυγμένο το οποίο αποψύχεται και θα πληρώσει περισσότερα για ένα καλό ψάρι αν έχει ενημερωθεί και σωστά γι' αυτό. Άρα είναι καλή αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μικρή κλίμακα αλία, πράγματι θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφοροποιημένο σύστημα για την αλία αυτή. Το έχω συζητήσει με το Συμβούλιο. Κάποια κράτη-μέλη, όχι πλειοψηφία όμως, το εξετάζουν το ζήτημα αυτό. Πώς να το θέσω. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένα με την προοπτική αυτή. Θα επιμείνουμε πάντως. Και θα επιμείνουμε διότι η παράκτεια, η μικρής κλίμακας... Ε, αλία ουσιαστικά έχει να κάνει με πιο αποδοτική αλία, πιο αποτελεσματική αλία. Είναι και πιο φιλική προς την απασχόληση η παράκτη αλία, η μικρή κλίμακα ε, αλία και δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης ε, στις παράκτιες κοινότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα, να διατηρηθεί η ζωή στις ακτές Κύριε Λεπάζ δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά ε, δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Θα πάμε και στη Σκοτία να βρούμε λύσεις για τις παράκτιες ε, περιοχές, για τη μικρή κλίμακα αλία. Θα μπορούσαμε ίσως να τους δώσουμε κάποια ξεχωριστά κονδύλια, να έχουμε μια ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό για τη χρηματοδότηση της παράκτης αλίας. Μπορούσαμε να τους δώσουμε κίνητρα επίσης για να συμμορφωθούν με τους κανόνες, διότι πρέπει να υπάρχουν εργαλεία, αλλιευτικά, ε, καινούργια δίχτυα κτλ. Θα τους δώσουμε λοιπόν περισσότερη χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό. Και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, τον τρόπο με τον οποίο αλλιεύουν, επιβάλλοντας αυστηρούς ελέγχους και κανόνες ε, στη μεγάλη κλίμακα, στη βιομηχανική αλλία όπως λέγεται. Έχω κάποια στοιχεία που θα μπορούσα να σας δώσω. Μέσα σε μια νύχτα μπορούν να ψαρέψουν ε, ε, όσο ψαρεύει όλη η μικρή αλή σε μια ολόκληρη περιοχή. Μιλώ για την βιομηχανική αλή. Τώρα, με την ηχθειοκαλλιέργεια. Το ίδιο πράγμα ισχύει. Δεν έχουμε επικεντρωθεί όσο θα έπρεπε στην, ε, στον τομέα αυτό. Θα υπάρχει όμως ξεχωριστή, ξεχωριστό κονδύλιο για τα σχέδια στον τομέα της ιδιακατοκαλλιέργειας και Θέλουμε πραγματικά να είναι βιώσιμος ο τομέας αυτός. Θέλουμε να υπάρχουν ε, κανόνες ε, για την ε, ευζοία των ηχθείων, για τη χρήση αντιβιωτικών κτλ. Υπάρχει ένα ζήτημα συμμόρφωσης, το παραδέχομαι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η συμμόρφωση είναι κάτι που πρέπει να συντονιστεί και με τις, σε επίπεδο κρατών μελών. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ε, βιολογική εκτιοκαλλιέργεια, είναι κάτι καινούργιο αυτό. Έχουμε ειδικού κανόνες, έχουμε ήδη λάβει αιτήματα χρηματοδότησης ε, σχεδίων για την ε, βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, τα κράτη-μέλη οι κυβερνήσει πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην μικρή κλίμακα αλία και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό σε ό,τι αφορά αυτές ε, τις ε, τράτες ε, και όλα τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και έχουν να κάνουν με τον βυθό. Έχουμε τον κανονισμό για τη Μεσόγειο Παραδείγματο χάρη που λέει ότι μετά από μία τριετή μεταβατική περίοδο πρέπει πλέον ο κανονισμός αυτός να εφαρμοστεί και άλλωστε ο κανονισμός είναι ιδιαίτερα φιλικός, ιδιαίτερα ευνοϊκός ε, για εκατοντάδες αλίες. Στην Ελλάδα για παράδειγμα 200-300 άτομα μόνο είναι αυτά τα οποία λεύουν σε μεγάλα σκάφη και όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα έρχονται να με βρουν για τα μεγάλα αυτά καΐκια που καταστρέφουν την Ποσειδονία και τα πάντα. Ε, ό,τι υπάρχει στο βυθό, διότι έχουν ε, στο πλευρό τους ε, τα λόμπι, έχουν δύναμη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση για τη μικρή κλίμακα. Άλλιας, για την όσπα τώρα, η τελευταία μου λέξη, Εκεί νομίζω είχαμε μια επιτυχία. Αρμόδιο είναι ο κ. Ποτότσνικ και οι υπηρεσίε του. Ήταν στην διάσκεψη τη ΩΣΠΑ που στέφτηκε από επιτυχία και τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν αυτές τις ε, περιοχές. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Ποτότσνικ και πραγματικά θέλουμε να δώσουμε κίνητρα, να παρακινήσουμε και άλλα κράτη-μέλη να ορίσουν προστατευμένες περιοχές. Επισκεφθήκαμε τη Γερμανία, έχουμε κάποια σχέδια εκεί αναφέρομαι και ε, στη Μεσόγειο. Τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. Φυσικά και πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη κτλ. κτλ. Δεν είναι δική μου η αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να σας πω εδώ. Ή μάλλον μπορώ να σας πω και πρέπει να σας πω ότι θα σεβαστώ την αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο αυτό που μπορούμε να κάνουμε όπως προείπα, είναι να χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό για την αλία IUU, την ε, παράνομη αδήλωτη άναρχη αλία. Διότι εάν ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, το προϊόν που αλλιεύουν και αν υπάρχει θέμα αλίας IUU, υπάρχει και ζήτημα επιστροφής κεφαλαίων των πληρωμών. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια να προχωρήσουμε σε τιμωρία, ιδίως αν πρέπει να τους τιμωρήσουμε όλους. Χρειαζόμαστε πραγματικά λοιπόν τη βοήθειά σας, τη βοήθεια των πολιτών για να πείσουμε τις κυβερνήσεις ε, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να δώσουν τα απαραίτητα μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very... Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι καταφέρατε να απαντήσετε σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Τουλάχιστον από σας θυμάμαι εγώ. Μπράβο σας. Μεγάλο επίτευγμα. Θα επανέλθουμε για το θέμα της Δυτικής Σαχάρας ε, πολύ σύντομα ούτως ή άλλως και θα ξαναπούμε με θέμα ακριβώς τη Δυτική Σαχάρα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Well, the next issue on the agenda is... Το επόμενο σημείο είναι η διασυνοριακή υγειονομική περίθευση Κυρία Γκοστέτ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουν παραμείνει λίγοι από εμά και είναι κρίμα γιατί το κείμενο είναι αρκετά, μάλλον ιδιαίτερο σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που είναι εδώ είναι πιο εργατικοί. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μια οδηγία που αφορά τα δικαιώματα των ασθενών για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ε, ασχολούμαστε από το 2004 ή αν όχι το 2004, σοβαρά το 2005 με την οδηγία. Πρέπει να σας πω ότι επήγει το θέμα αυτό, πρέπει να κλείσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα αρκετά πιεστικό, γιατί πιστεύουμε ότι απέναντι στους Ευρωπαίους ασθενείς έχουμε καθήκον να μην τους αφήσουμε εκτεθειμένους περισσότερο. Θα υπενθυμίσω το, το πλαίσιο πολύ σύντομα και εν συνεχεία θα περάσω στα βασικά σημεία, στα σημεία κλειδιά. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε μια συμφωνία επί Ισπανικής Προεδρίας, πολύ δύσκολη συμφωνία για την Ισπανική Προεδρία. Ήταν μια απρόσμενη επιτυχία από πλευράς της, που υποστηρίχθηκε από 20 κράτη-μέλη μόνο τρεις αντιθέσεις ε, υπήρξαν στο Συμβούλιο και μία αποχή. Η κοινή θέση του Συμβουλίου υιοθετήθηκε επίσημα στις 13 Σεπτεμβρίου και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Σεπτεμβρίου. Γιατί είναι δύσκολο το χρονοδιάγραμμα, γιατί καθυστέρησε το Συμβούλιο. Από την ε, συμφωνία αυτή επί Ισπανικής Προεδρίας μέχρι τη 13η Σεπτεμβρίου του 2010 πέρασε πολύς χρόνος χωρίς να γίνει τίποτε άλλο. Ποιο είναι ο στόχο αυτή τη οδηγία λοιπόν τώρα. Πρόκειται για τη διευκρίνηση των δικαιωμάτων των ασθενών όπω αναφέρονται και απαριθμούνται από το ΔΕΚ. Θα πρέπει να υπάρξει ασφάλεια δικαίου γενικώ σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη για του ίδιου του ασθενεί, αλλά και για τα κράτη-μέλη και τα εθνικά συστήματα κοινωνική περίθαλψης. Είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε την πρόσβαση και την ε, επιστροφή των ε, εξόδων υγειονομικής περίθαλψης, διασυνοριακός πώς, ε, σίγουρη περίθαλψη και ποιοτική περίθαλψη. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για, μεταξύ των κρατών μελών για τη υγειονομική αυτή περίθαλψη. Υπάρχει μια αρχή που πρέπει να υπενθυμίσουμε, είναι ότι το ΒΕΚ κάθε επανάληψη αναγνώρισε τα δικαιώματα των ασθενών και ο δικός μας ρόλος σήμερα είναι απλώς να κωδικοποιήσουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο αυτό που αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ούτω ώστε να ενδυναμώσουμε την ασφάλεια δικαίου και να εγγυηθούμε μία ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των δικαιωμάτων ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, για να μην υπάρχει αμφισημία, να υπενθυμίσω ότι με βάση τη συνθήκη οι κανόνες για την οργάνωση των ε, συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και αυτό δεν θα αμφισβητηθεί και δεν πρόκειται να συζητηθεί σε αυτό το κείμενο. Ποια είναι τα βασικά σημεία, τα σημεία κλειδιά του κειμένου. Καταρχάς, το κείμενο αφορά τους ασθενείς που έχουν ανάγκη και προβλήματα υγείας και όχι για τους ασθενείς που έχουν τα οικονομικά μέσα. Εδώ δεν θέλουμε να δεχτούμε και να προωθήσουμε τον ιατρικό τουρισμό. Τα βασικά σημεία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέραμε στην πρώτη ανάγνωση. Και αφορούν τα θέματα με το πεδίο εφαρμογή της οδηγία, τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των υγειονομικών εξόδων που παρέχονται διασυνοριακά και το θέμα της πρώτερης έγκρισης. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία τα οποία θα εξετάσουμε. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεκτικότητα ανάμεσα στη σημερινή οδηγία και στον κανονισμό 883 του 2004 που σκοπό είχε να εξορθολογήσει τους κανόνες και τις ε, διαδικασίες για το συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης των κρατών μελών, θα πρέπει αυτά τα δύο συστήματα ε, να συναθώνται σωστά. Όλοι γνωρίζουν αυτά τα νομοθετήματα, όλοι όσοι μετακινούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, καταρχάς η πρώτερη έγκριση η πρώτερη άδεια. Αυτό είναι κεφαλαιόδου σημασία σημείο. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάμωση τι είχαμε πει για αυτό το σημείο. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρώτερη έγκριση ε, για την νοσοκομιακή περίθαλψη, για την εξειδικευμένη περίθαλψη και για τη θεραπεία που παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή για τον γενικότερο πληθυσμό. Πρόκειται για την τροπολογία 55. Τώρα για το Συμβούλιο. Τι αποφάσισε το Συμβούλιο. Αποφάσισε να προσθέσει κάποιες προϋποθέσεις για την έγκριση και την εφαρμογή της. Κάποιες ανησυχίες που συνδέονται με την ποιότητα και την ασφάλεια. Άρθρο 8, παράγραφος 2 της περίθαλψης. Αυτό το κριτήριο, το οποίο προστίθεται από το Συμβούλιο, δεν είναι αποδεκτό. Γιατί θα επέτρεπε σε ανα πάσα στιγμή να αρνηθούμε την πρώτερη έγκριση χωρί κανένα δικαιολογητικό. Οποιοδήποτε κράτο μέλο θα μπορούσε να πει Α, δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, σίγουροι», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσει. Είναι αδιανόητο. Θα αντιμετωπίζαμε πάλι μια ασάφεια νομική, θα είχαμε εκ νέου προσφυγές στο ΔΕΚ και θα είχαμε εκ νέου αποφάσεις από το ΔΕΚ για το θέμα αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ένα σημείο επί του οποίου δεν υπαναχωρούμε. Εν συνεχεία, ποιε είναι οι προποθέσει για την πρώτερη έγκριση. Να υπενθυμίσω ότι για μα την πρώτη ανάγνωση είχαμε πει το εξή, ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ένα σύστημα πρώτερη έγκριση μόνο εάν η απουσία αυτής της πρώτη έγκρισης έθετε να αμφιβόλω την οικονομική ισορροπία του συστήματος κοινωνικής περίθαρψης και υγειονομική περίθαλψη του εν λόγω κρατου μέλου. Αυτή είναι η διάταξη που ψηφίσαμε στην πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο τι είπε. Δεν υπάρχει όρο, δεν υπάρχει προπόθεση. δεν υπάρχει θέση από πλευρά Συμβουλίου σε σχέση με αυτό το σημείο εδώ. Και εδώ θέλω να σε επιστήσω την προσοχή στο ότι η θέση του Συμβουλίου επανισάγει κάποιε νομικέ ασάφειε ε, που θα οδηγήσουν σε νέε προσφυγέ και που δεν είναι αποδεκτές με δεδομένη την ομολογία του δικαστηρίου. Και τώρα θέλω να πάω στους λόγους άρνησης της ε, πρώτερης αυτής έγκρισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απαριθμίσει τους λόγους άρνησης. Και εγώ τους αναφέρω αυτούς τους λόγους στην ε, τροπολογία μου υπαριθμών 59. Το Συμβούλιο προσθέτει και άλλους λόγους άρνησης της πρώτερης έγκρισης. Είναι μάλιστα ανοιχτό και μη εξαντλητικό ο κατάλογος αυτός. Το Συμβούλιο μιλάει ε, για αδύρυτου λόγους γενικού συμφέροντος. Αυτός ο, ο όρος είναι τόσο αόριστο, γενικός και αόριστος, που δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια άρνησης σαφή και εφαρμοστέα με τρόπο ομοιόμορφο στα κράτη-μέλη. Αλλιώ και εδώ θα δημιουργήσουμε τη δυνατότητα προσφυγών στο δικαστήριο και θα έχουμε προχωρήσει. Ούτε κατά κεραία. Σας εξήγησα τα σημεία από τον οποίο δεν επαναχωρούμε. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία, ίσως όχι τόσο σημαντικά όσο αυτά που σας ανέφερα ήδη. Να σας τονίσω το στοιχείο της ενημέρωσης του ασθενούς. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Πώς θα πρέπει να ενημερώνεται? Από τα εθνικά σημεία επαφής. Και εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το ρόλο αυτών των εθνικών σημείων επαφής. Αυτός ο ρόλος των σημείων επαφής είναι σημαντικός, γιατί χάρη σε αυτό ο ασθενής λαμβάνει τις απαραίτητες, χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες. Αυτό που ήθελε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, ήθελε αυτά τα εθνικά σημεία εφαρμογής να δικτυώνονται ούτως ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και επανάληψη των ιδίων διαδικασιών. Φανταστείτε, ένα ασθενή να πρέπει να πηγαίνει σε 27 διαφορετικά εθνικά σημεία επαφή να ψάχνει τι ίδιε πληροφορίε. Θα πρέπει το εθνικό σημείο επαφή του κάθε κράτους μέλους να δίνει τι καλύτερε πληροφορίε να πηγαίνει το ίδιο δηλαδή να ψάχνει τις πληροφορίες στα άλλα εθνικά σημεία επαφής, μέσω δηλαδή μιας δικτύωσης των εθνικών σημείων επαφής μεταξύ τους. Και εδώ έχουμε διαφορετική άποψη από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν θέλει να βάλει τόσες λεπτομέρειες αυτή τη διάταξη. Για μας τα σημεία επαφής πρέπει να, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητα για να ενημερώνουν καλύτερα τον ασθενή. Με γνώμονα μόνο το συμφέρον του. Καταθέτω λοιπόν και τα, τις τροπολογίες που υιοθετήσαμε για το σημείο αυτό στην πρώτη ανάγνωση. Για τα υπόλοιπα σημεία όπου υπάρχει διάσταση είναι η νομική βάση. Το Συμβούλιο λέει ότι πρέπει να υπάρχει διπλή νομική βάση σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά και το άρθρο ε, Δημόσια Υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούσε μόνο για την εσωτερική αγορά. Μπορούμε τελικά αρκετά εύκολα να δεχτούμε τη διπλή νομική βάση, γιατί δεν είναι απαράδεκτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον ύφαλο. Για το πεδίο εφαρμογή. Το Συμβούλιο θεωρεί προτείνει μάλλον να αποκλείσουμε την υγειονομική περίθαλψη μακράς διάρκειας από το πεδίο εφαρμογής, τη δωρεά οργάνων και την εκστρατεία εμβολιασμού. Και αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, δεδομένη τη εμπειρία που είχαμε το περασμένο χειμώνα. Καταλαβαίνουμε ότι το Συμβούλιο θέλει να αποκλείσει αυτού του είδου ε, την υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα όμως, οι ασθενεί που έχουν σπάνιες αρρώστιε θα πρέπει να υποφελούνται από μία επιστροφή, ακόμη και αν η θεραπεία δεν δίδεται με, βα στο δικό του κράτο μέλο. Υπάρχουν σπάνιε αρρώστιε για τι οποίε δεν υπάρχει θεραπεία σε κάποια κράτη-μέλη. Είναι αδιανόητο να τιμωρήσουμε δύο φορέ αυτού του ασθενεί. Από τη μία έχουν την ε, δύσκολη αυτή η σπάνια αρρώστια, δεν μπορεί να θεραπευτεί στη δική του χώρα, να του πούμε να πα σε μια άλλη χώρα, αλλά θα σου επιστρέφονται τα ιατρικά έξοδα. Όχι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτού του ασθενεί που πλήττονται από σπάνιε αρρώστιες. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή της προκαταβολής και την ε, εθελοντική πρώτερη έγκριση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν έχει δοθεί μια πρώτερη έγκριση, ο ασθενή θα πρέπει να πληρώσει καταρχήν μόνο το ποσό το οποίο θα έπρεπε να προκαταβάλει στη δική του χώρα. Το Συμβούλιο όμως λέει λέει τίποτα μάλλον, δεν λέει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ρήτρα. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα εδώ, γιατί είναι σημαντικό για τους ασθενείς. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αβεβαιότητα για την επιστροφή των εξόδων και τις προκαταβολές. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των ασθενών, ειδικά των λιγότερο εύπορων, που χωρίς αυτή τη διάταξη θα πέσουν θύματα διακρίσεων. Μην ξεχνάμε βέβαια, και δεν την ξεχνάω ούτε εγώ, την επικουρικότητα. Επίση, τι γίνεται με του συνταξιούχου που ζουν στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση. Το Συμβούλιο όμω ήθελε να συμπεριλάβει και του συνταξιούχου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το ιδιαίτερο αυτό σημείο. Είναι σημαντικό για κάποια κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να δεχτούμε το σημείο αυτό του Συμβουλίου. Και είναι σημαντικό να μην μπλοκάρουμε τη συμφωνία με το Συμβούλιο. Είναι λίγο ευαίσθητο και λεπτό αυτό το σημείο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας δημιουργήσει αντίρρηση στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τις διοντολογικές επιλογές, τις ηθικές επιλογές, είναι πολύ σημαντικό για κάποιους συναδέλφους. Η οδηγία, υπενθυμίζω, σέβεται και δεν θέτει να αμφιβόλο την ελευθερία που διαθέτει κάθε κράτος μέλος για να αποφασίσει το είδος της υγειονομική περίθαλψης θεωρεί το είδο τη ιδιωτική περίθαλψη που θεωρεί κατάλληλο. Καμία διάταξη τη οδηγία δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί με τρόπο ούτω ώστε να μειωθεί η δυνατότητα αυτή επιλογή για διοντολογικού λόγου που έχουν τα κράτη-μέλη. Θέλω λοιπόν να καθησυχάσω κάποιου κάποιου κάποιου συναδέλφου που του ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα σημεία, να μην ανησυχούν λοιπόν για αυτό το θέμα τη διοντολογία και τα ηθικά θέματα. Τέλο, να μιλήσω για τα ατομικέ ανάγκε. Ίσως υπάρχουν ιδιαίτερα έξοδα για την περίθαλψη των ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Φυσικά αυτό το επιπλέον κόστο θα πρέπει να επιστραφεί υπό κάποιε προποθέσει. Το πρόβλεψε αυτό το Κοινοβούλιο, αλλά το Συμβούλιο δεν δέχεται αυτό που πρόβλεψε το Κοινοβούλιο. Οι ειδικέ ανάγκε και οι αναπηρίε δεν αναφέρονται και αυτό δεν το δεχόμαστε. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Ασθενών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει να δημιουργηθεί μια τέτοια θέση για να διαχειριζόμαστε τις, τα παράπονα των ασθενών. Το Συμβούλιο δεν αναφέρει τη ρύθμιση αυτή, την πρόταση αυτή. Εγώ προσωπικά δεν είμαι πεπισμένη ότι είναι τόσο σημαντικό. Σας το λέω ειλικρινά, να αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαίο διαμεσολαβητή για τους ασθενείς. Θα ανοίξουμε τώρα ένα παραθυράκι για να δημιουργούμε επάπειρον διαμεσολαβητές επί διαμεσολαβητών. Δεν νομίζω ότι λύνονται τα θέματα με τη δημιουργία τέτοιων θέσεων. Σε ό,τι αφορά κάποιες περιοχές ε, δοκιμής, ιδίω στις διασυνοριακές περιοχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση αποφάσισε να προσδιορίσει τέτοιες περιοχές ε, δοκιμών, αν θέλετε, σε διασυνοριακές ε, ζώνες. Είναι πολύ σημαντικό για μας ε, το, το Συμβούλιο όμως δεν αναφέρει τίποτα επί αυτών. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε νέες εμπειρίες, συγκεκριμένες όμως, όπως συγκεκριμένα πειράματα. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει στις διαστηνοριακές περιοχές, μετά μπορεί να γενικευτεί και να είναι χρήσιμο. Επίσης, η ηλεκτρονική υγεία είναι πολύ σημαντική. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση ε, για την επιτροπολογία, το Συμβούλιο αντικαθιστά το σημείο αυτό με κατευθυντήριες γραμμές. Κατά την άποψή μου είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις, την ανάπτυξη που υπάρχει στην ηλεκτρονική υγεία. Το Συμβούλιο δεν δίνει σημασία στο σημείο αυτό και αγνοεί την ελπίδα που, γεννάει, που γεννάνε γενικά οι νέε τεχνολογίε. Λοιπόν, εγώ επανεισάγω όλε τι τροπολογίε τη πρώτη ανάγνωση. Η Ευρώπη έχει το δικαίωμα και το καθήκον να ε, μάθει από το, την τηλεφωνική υγεία, την ε, τηλεϊατρική και να εποφεληθούν ζώνες και περιοχές όπου η πρόσβαση στην υγεία και στην περίθαλψη είναι πολύ προβληματική, που δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί, αρκετοί γιατροί. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση ζητούσε μια πιο μεγάλη συμμετοχή των διαφερομένων, ειδικά σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση αυτών των τεχνολογιών υγεία. Οι διάφοροι εμπλεκόμενοι έχουν εμπειρία, έχουν τεχνογνωσία. Καλό είναι να εμπνευστούμε και να αξιολογήσουμε αυτές τις, ε, τεχνολογίες και πώς θα το κάνουμε αυτό, θα υποφεληθούμε από την εμπειρία τους. Επανισάγω λοιπόν τις ε, τροπολογίες ε, της πρώτης ανάγνωσης. Μαχόμαστε από το 2004, τόσο ώστε τα δικαιώματα των ασθενών, τα οποία αναγνωρίζει το ΔΕΚ, να παγιωθούν σε ένα νομοθετικό κείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπερασπιστεί τις θέσεις του, για, ειδικά σε ό,τι αφορά τα βασικά σημεία, τα σημεία κλειδιά. Αυτά τα θέματα ενδιαφέρουν τους πολίτες. Μιλάμε για την υγεία των πολιτών μας. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν. Αυτή τη στιγμή αυτοί που μπορούν να βασιστούν για να γνωριστούν τα δικαιώματά τους και να εφαρμοστούν πρέπει να προφύγουν αναγκαστικά στο δικαστήριο. Δεν μπορούμε να διαιωνίσουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ταράξουμε τα λιμνάζοντα ύδατα. Θα πρέπει πολύ γρήγορα γιατί ο χρόνος τρέχει και μετράει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια καλή δουλειά με συνεργασία, θα πρέπει γρήγορα να βρούμε μια λύση, υπερασπιζόμενοι προφανώς τα κρίσιμα σημεία απέναντι στο Συμβούλιο. Είμαι έτοιμη να σας ακούσω, ούτω ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση. Ευχαριστώ. Yeah. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε πολύ, Φρανσουάς Γκροστέτ, για την πολύ σημαντική αυτή νομοθετική προσπάθεια Εδώ το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο. Μπορεί μετά να δούμε τι κάνει το Συμβούλιο σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, άλλες θέλουν να κάνουν λίγα και άλλες είναι φιλικές προς εμάς. Θα ακούσουμε περισσότερα. Η Σκιώδης τώρα, η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το είπατε και εσείς κύριε Λάινεν ότι η έκθεση είναι σημαντική. Ένα θέμα που μας προβλημάτισε και μας και μας βασάνισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαίρω την Φρανσουάς Γκροστέτ για την έκθεση που είναι εξαιρετική, έντιμη σε σχέση με την πρώτη ανάγνωση και αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις μας, αλλά είναι και φιλόδοξη η έκθεση. Γνωρίζουμε την Φρανσουάζ, ξέρουμε ότι είναι φιλόδοξη και αυτό άλλωστε χαρακτηρίζει έναν ικανό πολιτικό. Διάβασα την έκθεση και προσωπικά θα μπορούσα όλα να τα υποστηρίξω. Αλλά μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα συμφωνήσουμε ώστε να μπορέσει πράγματι να τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή η, ε, το, η νομοθεσία. Το Συμβούλιο ε, δεν είναι τέλειο ως συνήθως στην κοινή θέση. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν διάβασα μια κοινή θέση του Συμβουλίου που να τη χειροκροτήσω και να πω τι ωραία που τα κάνατε. Ποτέ. Αυτό που σέβομαι στην κοινή θέση είναι ότι έγινε στο Συμβούλιο προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία και τα κατάφεραν. Η κοινή θέση δηλαδή αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Οπότε αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Γι' αυτό πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες προτεραιότητες θέτουμε εμείς που θα πλησιάσουμε το Συμβούλιο και που θέλουμε το, αντίστροφα το Συμβούλιο να πλησιάσει τις θέσεις μας. Δεν, μπορώ, δεν διεκδικώ τα ίδια δικαιώματα όπως η εισηγήτρια, ούτε θα μπω σε όλα τα θέματα. Μερικά θα θίξω. Ένα δεν είναι το σημαντικότερο βέβαια, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα θέμα που το έθεσα εγώ και αφορά τις σπάνιες ε, νόσους rare diseases. Πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της ύπαρξης σπάνιων νοσημάτων που δεν ε, προβλέπονται και δεν καλύπτονται οι δαπάνες, γιατί δεν υπάρχει η σε κάποια χώρα. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς παρόλα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάνε και να νοσηλευτούν εκεί που, όπου υπάρχει δυνατότητα. Και σίγουρα μπορούμε να τα βρούμε εδώ και με το Συμβούλιο, ώστε να βρεθεί μια καλή λύση. Ε, σε τρία από τα τέσσερα θέματα θα αναφερθώ. Η προτέρα άδεια για εξουσιοδότηση. Πριν κάνουμε την πρώτη ανάγνωση, ξέραμε ότι στις ομάδες, και στις ομάδες μας είχαμε κάνει πολύ εντατικές και δύσκολες πολλές φορές συζητήσεις. Προσπαθήσαμε όμως να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε. Η πρώτη ανάγνωση ήταν δύσκολη, αλλά τώρα μετά την κοινή θέση και αφού πέρασε και λίγος χρόνος, νομίζω ότι πιο εύκολα είναι τα πράγματα. Η προηγούμενη προτέρα εξουσιοδότηση είναι κάτι που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέει ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν το δικαίωμα και συμφωνώ κι εγώ ότι υπάρχει προτέρα εξουσιοδότηση ή άδεια. Το prior authorization, η προτέρα εξουσιοδότηση, δεν μπορεί όμως να είναι μέσον για να γίνονται καταχρήσεις και παραλογισμοί. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Ειλικρινή, Πρέπει όντω να υπάρχει επιθυμία για ορισμένε περιπτώσει να προβλέπεται προτέρα εξουσιοδότηση. Και από την κοινή θέση του Συμβουλίου αυτό δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο οπωσδήποτε χρειάζεται να δουλέψουμε εμείς περισσότερο. Βεβαίως ε, εκεί ε, το, στο Συμβούλιο είναι το ευάλωτο σημείο, το έθραυστο για το θέμα αυτό. Μετά, η όλη προβληματική των σημείων επαφής και των δικτύων. Η Φρανσουάς Γκροστέτε είπε επίσης ότι για τους ασθενείς είναι σημαντικό να έχουν κάποιους συνδέσμους, κάποια σημεία επαφής που να υπάρχουν εκεί και να είναι λειτουργικοί και να δίνουν πληροφορίες. Και τα δίκτυα όμως είναι σημαντικά ούτως ώστε να υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών για νοσηλίες, θεραπείες, ε, ε, βέλτιστες πρακτικές κλπ. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τα κράτη-μέλη την δυνατότητα να τα προσφέρουν όλα αυτά στους πολίτες τους. Όχι αύριο μεθαύριο, αλλά μέσω πρόθεσμα. Και ενδεχομένως θα βρούμε μια δυνατότητα να ορίσουμε το στόχο μας και να είμαστε και πιο ευέλικτοι χρονικά. Έπειτα, Δύο λόγια για το όλο πακέτο της ε, ανάκτησης των χρημάτων, της επιστροφής ή της ε, προκαταβολής ή της πληρωμής από το πριν. Μπορούμε να βρούμε σύστημα είτε με vouchers, με κάποια παραστατικά, κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη και στους ασθενείς να μην κάνουν πληρωμές μεγάλων ποσών από πριν και η επιστροφή που θα προβλέπετε να γίνεται γρήγορα. Ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη φοβούνται ότι αυτές οι επιστροφές των χρημάτων δεν λειτουργούν και υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά παραδείγματα κρατών μελών που περιμένουν πολύ ε, σε νοσοκομεία ατυχημάτων, που, ατυχήματα στις διακοπές ας πούμε. Περιμένουν πολύ μέχρι ότου ε, οι χώρες ε, προέλευσης ε, επιστρέψουν τα ποσά για τα νοσήλια και τις θεραπείες. Ε, αυτό μπορούμε όμως να το ρυθμίσουμε, να τους πούμε να φροντίσουν να γίνεται, να λειτουργεί το σύστημα επιστροφής. Τώρα η δεύτερη νομική βάση και... και εδώ μπορούμε να συνεννοηθούμε αν καταφέρομαι, και το λέω ιδιαίτερα αυτό προς την κατεύθυνση του Συμβουλίου, αν καταφέρομαι με την προτέρα εξουσιοδότηση και τους περιορισμούς ας πούμε που προβλέπετε, δηλαδή αυτά που είναι γραμμένα στο άρθρο 8, για να, να έχουμε ένα τροποποιημένο ορισμό. Νομίζω ότι στο άρθρο 8 πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πάλι αν ε, αυτή η μεγάλη περιορισμή που προβλέπει είναι όντως απαραίτητη και επίσης θα πρέπει να δούμε τους καταλόγους ε, που υπάρχουν για την πρώτερα εξουσιοδότηση. Η Φρανσουάζ Γροστέτ είπε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος. Αν λάβει απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θα αποφασίσει για επιμέρους υποθέσεις, αλλά για κακή διαχείριση, κακοδικία, μάλλον κακή εφαρμογή της νομοθεσίας. Και μετά θα προβλέψει και κυρώσεις και οικονομικές κυρώσεις κατά των κρατών μελών που δεν εφάρμοσαν την νομοθεσία. Ίσως ε, καλό είναι να το πούμε αυτό στο Συμβούλιο και να το συζητήσουν εκεί. Υπάρχουν κράτη-μέλη που λένε θα το ρισκάρουμε. Αλλά δεν θέλω να ελπίζω, δεν, θέλω να πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ε, είμαι αισιόδοξη. Πολλές συζητήσεις έγιναν. Υπάρχουν προοπτικές για ε, συμφωνία. Βέβαια και εγώ πολλές φορές ε, θέλω να ε, συμμετέχω στη συζητήση γιατί και στη δική μου την ομάδα υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις. Πάντως πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχία στη, μεταξύ εμείς με το Συμβούλιο. Είμαστε σε δεύτερη ανάγνωση, έχουμε τώρα στενά περιθώρια, άρα πρέπει να λειτουργήσουμε πολύ πειθαρχημένα και πάνω απ' όλα να θέλουμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εισηγήτρια ε, δόθηκαν που είναι και φιλόδοξη και ικανή. Αντώνια Παρβάνοβα. Να κοιτάμε και την ώρα γιατί δεν θα προλάβουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Φρανσουάς Γκρουστέτ για την έκθεση αυτή και μάλιστα είναι από τα πιο επίμαχα και περίπλοκα θέματα που πρόσφατα μας απασχόλησαν στο Κοινοβούλιο και όντως χρειάζεται όλη την υποστήριξη και τη συνεργασία μας για να βγούμε από μια κατάσταση που δυσκόλεψε τα τρία θεσμικά όργανα, Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και τα έφερε να διαμορφώ, τα έκανε να διαμορφώσουν αντιφατικές θέσεις. Όλα αυτά προέρχονται, βασίζονται ή έχουν σχέση με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν οριστικοποίησε τα οικονομικά θέματα και αν η δημόσια υγεία θα είναι μέρος της συνθήκης. Τώρα, πριν ξεκαθαριστούν αυτά τα θέματα, πάμε να προβλέψουμε εξαιρέσει για ασθενεί συγκεκριμένου που μπορεί να έχουν περισσότερα δικαιώματα από ό,τι εκείνοι σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να, είμαστε, να έχουμε κοινό μέτωπο για να προασπίσουμε όλοι μαζί τις προσδοκίες των ασθενών και το Συμβούλιο βέβαια έχει περισσότερα προβλήματα με την κρίση και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το θέμα της δημόσιας υγείας. Τρία θέματα θα αναφέρω ειδικότερα. Πρώτον, όπως είπα, οι ασθενείς και τα δικαιώματά τους και να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές της καθολικότητας, πρόσβαση ε, σε καλές υπηρεσίες υγείας, αλληλεγγύη στη ζωή όλων, σωστή κωδικοποίηση με βάση την ομολογία του δικαστηρίου και διατήρηση της οικονομικής και οργανωτικής βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, ούτως ώστε αφού εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, να μην τους εκθέσουμε σε μεγαλύτερες δυσκολίες από τις τωρινές. Τώρα, για τα συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται, ειδικότερα εθνικά σημεία επαφής άρθρο 6 της θέσης του Συμβουλίου, συμφωνούμε απόλυτα με την εισηγήτρια που δίνει πάλι ε, καλύτερο περιεχόμενο στη διάταξη και αν μιλάμε για δικαιώματα ασθενών πρέπει να φροντίσουμε ότι θα είναι ξεκάθαρα διατυπωμένα και θα τα γνωρίζουν. Ο ρόλος των εθνικών σημείων επαφής θα πρέπει να οριστεί όσο γίνεται πιο επακριβώς. Τώρα, για την επιστροφή των δαπανών άρθρο 7, όποια και να είναι η απόφαση, η απόφαση αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί ανισότητες και θα βοηθάει τα διαφορετικά συστήματα υγείας των κρατών μελών που είναι διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι ασθενείς θα εκτεθούν σε μεγαλύτερες δυσκολίες και μόνο με το ταξίδι στο εξωτερικό, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε το δικαίωμα, το δικαίωμα αυτό να μην τους επιβαρύνει οικονομικά κατά την άσκησή του όταν το ασκούν. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκρίσιμο ή ενιαίο σύστημα για όλους τους ασθενείς. Προτεραιότητες, άρθρο 8 της ε, θέσης του Συμβουλίου, συμφωνούμε απόλυτα με την προσέγγιση της εισηγήτρια και πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμείνει στο, θέμα αυτό. Τώρα, για την εξαίρεση ε, όταν έχουν σπάνιες νόσους από την πρώτερη εξουσιοδότηση ή άδεια, απόκτηση είναι λίγο παράδοξη αυτή η κατάσταση κατά την οποία προσπαθεί η Κομισιόν να αντιδράσει σωστά και έγκαιρα στις απαιτήσει που υπάρχουν από την πλευρά των, και τις ανάγκες των ασθενών και των οργανώσεων που έχουν σπάνια νοσήματα. Αλλά δεν είναι καλή θέση εδώ γιατί αυτή είναι η μόνη εξαίρεση στην οδηγία που θα δημιουργήσει ανισότητες μάλλον και διακρίσεις πάνω στη βάση των ασθενειών, αν είναι σπάνια ή όχι. Και κράτη, σε κάποια μπορεί να μην υπάρχουν ασθενείς με σπάνια νοσήματα. Συνολικά όμως είναι 11 εκατομμύρια οι ασθενείς στην Ευρώπη με σπάνια νοσήματα. Φαντάζεστε τι ταξίδια μπορεί να λάβουν χώρα αν δεν προσέξουμε ιδιαίτερα τις εξαιρέσεις αυτές. Και πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα και να δούμε αν υιοθετήσουμε αυτή την οργανωτική προσέγγιση, ενδεχομένως και άλλες ομάδες ασθενών, μικρότερες σε μέγεθος, θα θεωρήσουν ότι καλύπτονται. Τώρα για την ηλεκτρονική υγεία, το άρθρο 13, αυτή η οδηγία δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε αποτελεσματικότητα, και καινοτομία, ασφάλεια. Ε, δεν θα μακρηγορήσω γιατί είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Μία ερώτηση για την αξιολόγηση της ε, τεχνολογίας υγείας. Ιδιαίτερα η συγγύητρια στην ε, τροπολογία 88 προτείνει παροχή πληροφοριών σχετικά με τη σχετική αποτελεσματικότητα και στην τεχνολογία της υγείας. Έφικαση, αποτελεσματικότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε σχέση με την τεχνολογία πριν. Α, efficacy λέγεται η αποτελεσματικότητα πριν η τεχνολογία κυκλοφορεί στην αγορά και effectiveness αφού, όπως κρίνεται η αποτελεσματικότητα, αφού κυκλοφορεί στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πολύ μεγάλο αυτό φάκελο με όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και όπως ε, και η συνάδελφος Ροτ Μπέρεντ, ε, συμφωνώ και εγώ ότι θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία να εξασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο θα προσεγγίσει το Κοινοβούλιο στη δεύτερη ανάγνωση. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, τρία ακόμη μείζωνα ζητήματα από δική μας πλευράς για τα οποία θεωρούμε ότι καλό είναι να το επεξεργαστούμε ακόμη περισσότερο σε σχέση με αυτό που είπε και η συγγήτρια. Για τα λοιπά σημεία είμαι σύμφωνη, μπορώ να σύμφωνος και μπορώ να υποστηρίξω ότι είναι η συγγήτρια. Νομίζω ότι πολύ καλά επαναλαμβάνει τα σημαντικά για μας σημεία της πρώτης ανάγνωσης συγγήτρια. Λοιπόν, ποια είναι αυτά που πρέπει να συζητηθούν ακόμη στο Κοινοβούλιο από αυτά τα τρία που είπα. Πρώτον, η πρώτερη έγκριση. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι αν μιλάμε για λόγους ε, άρνησης της πρώτερης έγκρισης, αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε έναν πλήρη κατάλογο. Το Συμβούλιο δεν ακολούθησε σωστή διαδικασία, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε στο Κοινοβούλιο, γιατί ο κατάλογος δεν ήταν εξατλικός, δεν ήταν πλήρης. Τώρα, η συγκέντρια δεν αναφέρει λόγους άρνησης της επιστροφής ε, των δαπανών. Νομίζω ότι εμείς ε, θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το ζήτημα ως Κοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι Υπάρχουν λόγοι γενικού ενδιαφέροντος, παραδείγματο χάρη υπονόμευση της οικονομικής ισορροπίας του δημοσιονομικού συστήματος. Αυτό είναι ένας λόγος για να αρνηθεί κανείς την επιστροφή δαπανών. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω από την εισηγητρία λέει αν κάποιος είναι ασθενής και θέλει να λάβει μια θεραπεία σε μια άλλη χώρα θα πρέπει να εφαρμόσει, να πρέπει να τηρήσει τους κανόνες του κράτου σε αυτού. Αν χρειάζεται λοιπόν προκαταβολή, ακόμη και αν ο ασθενής είναι από ένα άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να καταβάλει την προκαταβολή αυτή. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και στο κράτος ε, με προορισμού. Νομίζω θα πρέπει λίγο να αλλάξει η στάση του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις ε, σπάνιες ασθένειες τώρα, το τρίτο ζήτημα που θέλω να σχολιάσω, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να επεκταθούμε λίγο. Η θέση του Συμβουλίου ε, δεν είναι παραδεκτή, δεν αναφέρεται σπάνιες ασθένειες, αλλά το να δώσουμε και μία ενλευκό εξαίρεση από την πρώτερη έγκριση είναι κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνο και νομίζω ότι συμφωνούν, ε, συμφωνεί και ο συνάδελφος από τους φιλελευθέρους. Έχουμε πρόβλημα στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό. Όταν ε, έχουμε να κάνουμε με μια σπάνια ασθένεια, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, αν για κάποιο κράτος μέλος κρίνεται σκόπιμο, να μπορεί να υπάρξει άρνηση Τη πρώτερη έγκριση. Αυτά τα τρία λοιπόν ζητήματα νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν ω Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να κινηθούμε λίγο, θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο, αλλά σίγουρα μπορούμε να εμείνουμε σε αυτή την πολύ ισχυρή θέση και έτσι να κερδίσουμε και στην δεύτερη ανάγνωση αυτά τα οποία θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της. Η όλη θεματολογία είναι σύνθετη και ευρύτατη. Εγώ θα ε, μιλήσω για κάποιες αρχές. Υπενθυμίζω ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τη νομική ασφάλεια των πολιτών, όλων των πολιτών, όχι μόνο εκείνων που ενημερώνονται καλύτερα. Θέλουμε να μην διαταράξουμε τη νομική ασφάλεια των συστημάτων. Τώρα για την πρόσβαση στις πληροφορίες θέλουμε όσοι, όλοι να μπορούν να έχουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αν χρειάζεται και πρέπει να είναι προσβάσιμες και εύληπτες οι πληροφορίες ακόμα και για άτομα ανάπηρα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις άλλες τις πληροφορίες για όλο τον πληθυσμό. Είμαστε στον 21ο αιώνα και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε όλες ε, οι ηλεκτρονικές μορφές να είναι προσπελάσιμες για την πληροφόρηση. Γι' αυτό ε, θα υποβάλω σχετικές ε, τροπολογίες. Επίσης, μία παράμετρος της υγειονομικής περιθαλψής είναι η ποιότητα και η ασφάλεια της φροντίδας που παρέχεται παντού. Πρόκειται πάνω απ' όλα για τη συνέχεια της παροχής αυτής της φροντίδας. Η συνέχεια επηρεάζεται και από την ε, πληροφόρηση και σε ηλεκτρονική μορφή που είναι πληροφορίες που μπορούμε εύκολα να ταξινομήσουμε και να διοχετεύσουμε παραπέρα. Προϋπόθεση για την διαβίβαση είναι η διαλειτουργικότητα, οπότε ο μεμονωμένος χρήστης να συνεννοείται με τους άλλους. Και στην ε, υγειονομική περίθαλψη χρειάζεται ενημέρωση των ασθενών. Όσοι θα επιθυμούν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη πρέπει να ε, έχουν το δικαίωμα να ε, ενημερώνουν και όσοι πήγαν στο εξωτερικό θα πρέπει να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και την, ε, τις πληροφορίες που αποκόμισαν. Και ε, αν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή πληροφορίες, τότε ο, δικαιο, ο κάθε ασθενής θα πρέπει να μπορεί να παίρνει τις πληροφορίες αυτές και να τις χρησιμοποιεί. Είναι σημαντική λοιπόν η διαλειτουργικότητα στις πληροφορίες. Πώς θα καταφέρομαι να είναι διαλειτουργικές. Η διαλειτουργικότητα είναι η προϋπόθεση για την ποιότητα της περίθαλψης. Και είναι και προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών να ρυθμίσουν το θέμα αυτό το ταχύτερο δυνατόν με κανόνες που θα εξασφαλίζουν διαλειτουργικά συστήματα. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν κοινού κανόνες ακόμη. Οπότε η Κομισιόν θα πρέπει να ε, δημιουργήσει αυτούς τους κανόνες. Επίσης κανόνες ε, ταυτοποίησης και έγκρισης. Πρέπει να δούμε ακόμα και τον ορισμό ε, της υγείας. Θέλουμε οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν φάρμακα σε όλες τις χώρες. Χρειάζεται λοιπόν και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τα συστήματα συνταγογράφησης πρέπει να είναι συμβατά για να γίνει αυτό, για να ελέγχεται η γνησιότητα της συνταγής. Χρειάζεται δυνατότητα επαφής μεταξύ του γιατρού που συνταγογράφησε και του φαρμακοποιού, ο οποίος θα το δώσει. Ε, μιλάμε εδώ για πληροφορίες και εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών υγείας. Χρειάζεται εδώ ανταλλαγή πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι ερευνητές και η βιομηχανία και οι γιατροί Τέλος για την ηλεκτρονική υγεία 20 δευτερόλεπτα. Με την προτέρα έγκριση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο και ηλεκτρονική υγεία. Εδώ έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών. Εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαι με αυτό το θέμα και θα ήθελα να δημιουργηθεί μια άτυπη ομάδα εργασίας για αυτό το θέμα. Η Επίτροπος Ρέντινγκ άλλωστε εξεδήλωσε ενδιαφέρον να επακοινωνήσει με μια τέτοια ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η σκιώδηση. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Μάξιμουμ τρία λεπτά δεν θα προλάβουμε. Που αν όχι, ο κύριος Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Έχω σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του κειμένου. Γιατί? Από τη μία δίκαιο είναι να επιτρέψουμε στους ασθενείς να κινούνται ελεύθερα και να υποφελούνται από η υγειονομική περίθαλψη που χορηγείται σε άλλα κράτη, αλλά όχι στη χώρα τους, Φερρυπίν. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ένα σύστημα που εγγυάται σε χώρες που λόγω ευθύνη άλλων κρατών μελών ε, κατακλείζονται από άτομα, ας πούμε, ασθενείς άλλων κρατών μελών, επειδή, ας πούμε, κάποιες θεραπείες δεν υπάρχουν στο, ε, αρχικό κράτος μέλος, ε, δεν προστατεύονται. Εδώ μιλάμε απλώς για ελευθερία μετακίνησης των πολιτών, των ασθενών. Μόνο και μόνο για να μειωθούν, λέει, ας πούμε, κάποιες λίστες αναμονής, δυνατότητα μετα... μετακίνησης από το ένα κράτος μέλος α στο β. Ας πούμε, έχουμε δύο κράτη-μέλη, το α και το β. Κάθε κράτος είναι κυρίαρχο στο τι θεραπείες θα προσφέρει και τι κόστος θα έχει κάθε θεραπεία. Έχουμε το α και το αβ, ας πούμε, κράτος μέλος. Το αβ δεν έχει ε, καλή θεραπεία. Το Β έχει όμως καλή θεραπεία. Αν μετακινούνται εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς από το Α στο Β, πώς θα μπορέσει αυτό το κράτος Β που πολιορκείται από άτομα τα οποία έχουν ανάγκη από θεραπεία, από θέσεις ε, νοσοκομεία, από ιατρικό εξοπλισμό, αλλά πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, οικονομικός πώς. Στο κείμενο λέμε ότι το τμήμα που επιστρέφεται από το κράτος από το οποίο προέρχεται ο ασθενής δεν είναι εκείνο όπου θα δοθεί η θεραπεία στον ασθενή. Μπορεί, δηλαδή, ανάμεσα στα α και β δεν έχουμε... Δεν μετακινούμαστε μόνο από το α στο β. Μπορεί να μετακινηθεί κάποιος σε ένα τρίτο κράτος μέλος. Ας πούμε, ε, στην Ιταλία έχουμε την ε, περιοχή του Βένετο. Αν αύριο μεθαύριο διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπει ένα κράτο που δεν έχει καλή οικονομική υπέρφλεψη, ε, αν φτάσουν ας πούμε 100.000 ασθενεί από την ε, τρίτη χώρα ε, στο Βένετο για να θεραπευθούν, τι γίνεται. Δεν καταραίει το υγειονομικό σύστημα του Βένετο. Τι εγγυήσει υπάρχουν για την περιοχή αυτή του Βένετο. Έτσι. Με την τροπολογία σας, κυρία εισηγήτρια, θα καταργήσετε τη μοναδική ρήτρα διαφύλαξης που έχει βάλει το Συμβούλιο στο κείμενο, μιλάω για το άρθρο 7-9, όπου λέει για λόγους ύψης του γενικού συμφέροντος, σας τελείωσε ο χρόνος, τρία λεφτά είχαμε πει. Πέντε νόμιζα, λέει ο κύριος Ρώση. Όχι, όχι, τρία. Ε, Πέτα Λίζε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γκροστέτ. Αυτή είναι η σημαντικότερη έκθεση στον τομέα της υγείας και με μεγάλη αφοσίωση και ε, γνώση συνέχισε το έργο του κυρίου Μπόις. Θα ήθελα να πω μετά τον κύριο Ρώση ότι δυστυχώς συχνότατα εντοπίζομαι τα προβλήματα από τη διασυνοριακή περίθαλψη. Ακούω όπως γιατρούς που χαίρονται όταν ασθενείς ε, μπορέσουν να πάνε στη Γερμανία μετά από τόσο καιρό αναμονής. Όχι, δεν θα κατακλειστούμε, δεν το φοβόμαστε αυτό. Το 1 τρίτο βέβαια των δαπανών επιστρέφεται και αυτό δεν συνάδει ούτε με την πρόταση της Κομισιόν ούτε με την πρόταση της κυρίας Γκροστέτ. Βεβαίως ε, θα επιστρέφονται οι δαπάνες, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε επικοδομητικά προς το συμφέρον των ασθενών και πιστεύω ότι όλοι θα ωφεληθούν. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και το ρίσκο δεν πρέπει να το δραματοποιούμε τόσο πολύ όπως κάνουμε κάποια φορά. Εγώ υποστηρίζω την έκθεση της κυρίας Κροστέτ και σε τρία σημεία θέλω ε, να ε, τονίσω την ανάγκη αλλαγής της κοινή θέση. Πολλά είπαμε για τις σπάνιες ε, νόσους. Αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 80 της Φρανσουάζ, όπου εδώ και το Συμβούλιο ήθελε να μας προσεγγίσει, ώστε να αναφερθούν τουλάχιστον, να γίνει μνήα των σπανίων νοσημάτων. Τώρα, αν θα περάσουν οι 47 με τη σειρά αυτή, αλλά πρέπει να δώσουμε μάχη ούτω ώστε οι σπάνιες παθήσεις των ασθενών να αντιμετωπίζονται και να τους ε, ε, βοηθήσουμε λίγο αν δεν προβλέπεται η επιστροφή δαπανών σε ορισμένα κράτη-μέλη. Γιατί καμιά φορά είναι τόσο σπάνιες οι παθήσεις που ναι δεν υπάρχει η ε, νόσος, γιατί η Ντάγμα Ροτμπέρντ είπε ότι δεν υπάρχει η νόσος. Όχι δεν υπάρχει νόσος, ήταν λάψους της Ντάγμαρ. Ε, υπάρχει η νόσος, δεν υπάρχει η θεραπεία παντού. Είμαι ευγνώμων γιατί οι 1 και 5 επανακατατέθηκαν για την ε, ε, δεοντολογία και τη διαφορά και είμαι και ευγνώμων για την 53 το θέμα του Βάουτσερ, Ξέρω ότι είναι δύσκολο και στην ομάδα μας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά ως άμεσα εκλεγμένοι πολίτες πρέπει να θεωρούμε σημαντικό να μην κολλήσουν στα χρήματα οι ασθενείς βέβαια. Δεν είναι καθόλου ωραίο αν δεν επιστρέφουν τις δαπάνες τόσο γρήγορα ε, τα ταμεία. Αλλά το χειρότερο είναι να, πάρει προκατα... να δώσει προκαταβολή ασθενή και να μην πάρει τα χρήματα. Άρα η 53 είναι η σωστή προσέγγιση και πρέπει να βάλουμε πλάτη στη Φρανσουάζ στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ιολάντα. Ευχαριστώ. Ομολογώ. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι η έκθεση Γκροστέτ είναι υποδειγματική. Ε, είμαστε ευγνώμονες για την εργασία σας, γιατί όλοι μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη θέση και είμαι πολύ ικανοποιημένη για το γεγονός ότι ε, κατέληξε σε μια συμβαστική λύση, όχι απόλυτα ικανοποιητική, το Συμβούλιο, αλλά πάντως ε, έκανε ένα βήμα προς την κατεύθυνσή μας για να λύσει προβλήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Πολλές φορές συζητήθηκε σε όλα τα κράτη το θέμα αυτό και στο επίπεδο του Συμβουλίου, αλλά και στο Κοινοβούλιο. Στην πρώτη ανάγνωση ως γνωστόν υπήρχαν ε, διαφορές. Ξέρω ότι η συμβαστική λύση αυτή δεν είναι εύκολη και ούτε είναι δυνατόν να μείνουν ικανοποιημένοι όλοι. Πάντως διαπιστώνουμε ότι αν καταφέρουμε να επεξεργαστούμε μια τέτοια συμβιβαστική λύση, ώστε οι βασικές προϋποθέσεις για τη βοήθεια των ασθενών θα είναι καταγεγραμμένες και αποδεκτές από όλους, τότε αυτό θα είναι μεγάλο γεγονός για το κοινοβούλιο μας. Αναμφίβολα, η οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών είναι αναγκαία κατεπηγόντως και ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. αν στη χώρα τους δεν μπορούν να έχουν γρήγορη και πλήρη θεραπεία. Αυτή η διατύπωση είναι σίγουρα λύση καλή, η οποία ε, επηρεάζει θετικά τα δικαιώματα των ασθενών. Έτσι, η περίθαλψη των ασθενών βελτιώνεται σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία ενιαίου συστήματος, γιατί κάθε κράτος μέλος έχει το σύστημά του. Εδώ πρόκειται μάλλον για μια διεύρυνση των δυνατοτήτων ε, θεραπείας και της πρόσβασης σε θεραπεία σε άλλα κράτη. Και η Πολωνία μεταξύ άλλων ε, είχε προβλήματα με αυτή την οδηγία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον τουρισμό νοσηλειών. Δεν το φοβούμε θα πια αυτό, ε, εγώ δεν το φοβούμε πια, διότι εδώ υπάρχει κάποιο εμπόδιο ότι το κράτος μέλος θα επομιστεί τις δαπάνες που θα λάβουν χώρα και προβλέπονται για τη συγκεκριμένη θεραπεία σε αυτό το κράτος μέλος. Αν αποφασίσει ένας ασθενής να επιλέξει άλλο κράτος και να πάει να κάνει εκεί τη θεραπεία του, τότε ενδεχομένως θα πρέπει και εκείνος να πληρώσει από την τσέπη του κάτι. Ε, δεν είναι τόσο γενικό το πρόβλημα πολλές υπηρεσίες ε, υποτιμώνται πολλές φορές στον τομέα της υγείας, ε, όχι στη Γερμανία, αλλά ε, σε χώρες όπου θεωρείται το σύστημα καλό όπως στη Γερμανία δεν κατακλείζονται. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ευνηδίως χρειάζεται κατεπηγόντως διασυνοριακή περίθαλψη και τότε είναι καλό να υπάρχει. Κριστίνα Γκουτιέρετ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την Φρανσουάζ Γκροστέτ ε, στο 99%. Και με την Τάγμαρ συμφωνώ και νομίζω ότι είναι σωστή η εστίαση της έκθεσης. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Ισπανία δημιούργησε την ε, μειοψηφία ε, της, που μπλοκάρει ουσιαστικά τις εξελίξεις και αυτή είναι που ουσιαστικά ξέμπλεξε, απέσυρε αυτή τη μειοψηφία. Όταν Μία ε, χώρα στέλνει έναν ε, ασθενή, ορίζει τι κοστίζει και η άλλη χώρα που δέχεται τον ασθενή ε, παρέχει την αγωγή, τη θεραπευτική περίθαλψη. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε. Σιγά σιγά θα προσεγγίσουμε μια χώρα την άλλη. Στον καρκίνο μια χώρα χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, άλλη όχι, παραδείγματος χάρη με την ακριβή χημειοθεραπεία. Σε πολλές χώρες γυναίκες ε, πάνω από τα 60-65 δεν έχουν το δικαίωμα της ακριβής αυτής θεραπείας, της χημεθεραπείας δηλαδή. Δεν αναφέρονται στα στατιστικά στοιχεία, αλλά εμείς είχαμε ε, ουσιαστικά ιατρικό τουρισμό. Ήρθαν πάρα πολλοί ασθενείς που δεν μπορούσαν να λάβουν θεραπεία στις χώρες τους ε, και υπάρχουν μεν κάτοικοι οι οποίοι δεν πλήρωναν, δεν πλήρωναν φόρους, αλλά ζούσαν. ζούσαν. Και αυτό το θέμα ε, πραγματικά έχει τεθεί, πρέπει να τεθεί. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί Βρετανοί, Γερμανοί, Πικοί, ε, είναι στην Ισπανία, αλλά χωρίς να πάρουν ε, την άδεια παραμονή, γιατί αν πέθαινε ο σύντροφο, παραδείγματο χάρη, δεν μπορούσαν να ενταχθούν ε, ξανά στη χώρα και γι' αυτό και δεν ε, έπαιρναν την άδεια παραμονή στην Ισπανία. Δεν μπορεί κάποιο να πει ότι πάω στη χώρα μου και ανακτώ όλα τα δικαιώματά μου. Σε άλλε περιπτώσει μπορεί. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για του ανθρώπου που ζουν σε μια άλλη χώρα από τη χώρα ε, τη καταγωγή του. Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχει ένας ρόλος για τον οποίο αντιτάχθηκε η Ισπανία χρειαζόταν τους δύο νομικούς πυλώνες, όχι έναν μόνο. Η χώρα υποδοχή στην πρώτη εκδοχή, η χώρα υποδοχή του ασθενούς δεν μπορούσε να επιβάλλει περιορισμούς ε, και ο ασθενής επέλεγε το νοσοκομείο. Φυσικά θα πάνε όλοι στο πιο ακριβό και καλό ε, νοσοκομείο της Μαδρίτης ή τέλος πάντων αν το καλύτερο καρδιολογικό είναι στην θα πάνε εκεί το αντίστοιχο αλλά το κράτος υποδοχής έχει και κάποια δικαιώματα να πει εγώ μπορώ να δεχθώ παραδείγματο χάρη 90, 150 χειρουργές επεμβάσεις στο χρόνο. Πρέπει να μπορεί να βάλει κάποια όρια. Μόνο αν δρομολογηθούν κάποια πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα άρουμε και εμείς τις ενστάσεις μας και θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Από την άλλη πλευρά σίγουρα καλύπτεται ένα νομικό κενό γιατί θα περιοριστεί ο ιατρικός τουρισμός. Για την περίπτωση της ε, Βενετίας χάρη. Πράγματι, σήμερα η απειλή είναι μεγαλύτερη που δεν είναι ρυθμισμένο και οργανωμένο το σύστημα. Όταν θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, διακόπτει ο πρόεδρος, διακόπτει. Συγγνώμη σας διέκοψα, Γιάννος Άντα, επόμενος. Τρεις ομιλητές ε, απομένουν. Δυστυχώς μας τελειώνει ο χρόνος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αξιέπαινο πως η κυρία Γκροστέτ τη θέση του Συμβουλίου την ε, αμφισβήτησε αποφασιστικά και με συνέπεια. Τρία θέματα ε, πρέπει να πω. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Η πρόταση της ε, είναι πολύ πιο σαφής και ξεκάθαρη διατύπωση από εκείνη του Συμβουλίου. Να την υποστηρίξουμε επίσης για το σύστημα ενημέρωσης. και το θέμα του δικαιώματος για ενημέρωση των ασθενών. Υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος που δεν τονίστηκε μέχρι τώρα. Δηλαδή, οι υπηρεσίες υγείας, εκείνοι που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας πρέπει να ξέρουν πολύ καλά και εκείνοι ποιος είναι ασφαλισμένος και ποιος όχι. Για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή. Επίσης, η υπηρεσίες ε, καθάρισης των λογαριασμών. Το σύστημα, ανεξάρτητα από το που θα γίνει, θα πρέπει να λειτουργεί με επαγγελματισμό, ταχύτητα, αξιοπιστία. Λοιπόν, και αυτό θα πρέπει να ε, μιλισμονηθεί. Επίσης, ε, ε, δεν ισχύει παντού το ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα αποφεύγονται προβλήματα με τη μετατροπή. Επίσης, με ειδική πλειοψηφία πρέπει να ληφθεί η απόφαση μετά τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, αν θέλουμε να περάσουν οι προτάσεις μας. Προετοιμάζοντας τις αποφάσεις, τις συνεδριάσεις των Επιτροπών, αλλά και στην Ολομέλεια, θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό το θέμα αυτό. Αν δεν έχουμε την ειδική πλειοψηφία, μπορεί να χάσουμε. Επίσης υπάρχουν και άλλες αντιφάσεις ε, προβλήματα που ε, αντιμετωπίζονται μέσα από τις τροπολογίες. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τώρα μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που υπήρχε από παλιά. Στα Ουγγρικά ε, λέμε μια παροιμία ε, να, να προσέξουμε να μην έχουμε το όρος όρο έτσι και μην. Linda um, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επί της ουσίας, ό,τι αφορά την πρώτη έγκριση, συμφωνώ με την Ντάγμαρ ε, ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη θέση του Συμβουλίου για να καταλήξουμε σε συμφωνία ένα ακανθόδη ζήτημα. Ε, σωστά λέει η κυρία Γκροστέτ ότι είναι λίγο υπερβολικά ανοιχτό αυτός ο κατάλογος, αλλά τελικά ε, πρέπει να αποφασίσουμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Η πρώτη έγκριση, ναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Για τις πάνες ασθένειες τώρα, ρωτώ την Επιτροπή, αυτός ο νέος νόμος πώς σχετίζεται με τον κανονισμό 883. Γιατί συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορούν ε, υπό το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης ε, οι άνθρωποι να πάνε στο εξωτερικό ε, και να καλυφθεί πλήρως το κόστος, να καλυφθούν πλήρως οι δαπάνες. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με την πρώτερη άγκριση και τις σπάνιες ασθένειες, γιατί είχαμε περιπτώσεις ε, που είχαν κάποιες ε, ε, περιπτώσεις που άνθρωποι απεγνωσμένοι πραγματικά ένας με σκλήρινση κατά και που είχε χαλάσει χιλιάδες απεγνωσμένος έφυγε και πήγε κάπου αλλού λοιπόν πρέπει να το ελέγξουμε γιατί ο κόσμος που είναι άρρωστος πραγματικά είναι απελπισμένος καλό είναι λοιπόν να έχουμε έναν κανονισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης για το θέμα αυτό θέλω να υποστηρίξω τώρα την εισηγήτρια στο ζήτημα της ανταλλαγής ε, πληροφοριών ε, για ε, κακές πρακτικές. Θα πρέπει οι ρυθμιστές, οι αρχές να γνωρίζουν τι γίνεται με γιατρούς ή επαγγελματίες του κλάδου της υγείας οι οποίοι ε, έχουν κάποιες καταχρηστικές πρακτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ε, καταλαβαίνω ποιο είναι το ζήτημα με την ισότητα πληρωμών Έχουμε ένα σύστημα για την αποζημίωση, την επιστροφή για την κάρτα υγείας. Ξέρουμε ότι επιστρέφονται μετά από χρόνια ε, τα ποσά αυτά. Πώς ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να δεχθεί έναν ασθενή όταν η κυβέρνηση που υποτίθεται να, πληρώ, να πληρώσει ε, πληρώνει μετά από χρόνια. Πόσα χρόνια πια να περιμένει αυτό το νοσοκομείο. Εσείς ουσιαστικά θέλετε να σταματήσετε την μετακίνηση των ασθενών και όχι να τη διευκολύνετε. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, φυσικά και δεν μπορούμε να έχουμε έναν διαμεσολαβητή, δεν μπορούμε να δημιουργούμε τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια για κάθε ζήτημα. Σε ό,τι αφορά όμως τα σημεία επαφής, ναι, πρέπει να υπάρχουν σημεία επαφή τα οποία θα αναλογούν, θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που μετακινούνται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τι κυβερνήσει να δημιουργήσουν σημεία επαφή που θα δουν πληροφορίε για θεραπείε στο εξωτερικό. Αυτό ούτε για την ίδια του τη χώρα δεν μπορούν να το κάνουν προ το παρόν θέλω να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πόσα άτομα μιλάμε. Πόσοι το θέλουν αυτό. Και το τελευταίο σχόλιο. Για ένα συνάλφο που μίλησε για εξοπλισμό, για συνταγηγογραφήσεις, για ένα τεράστιο σύστημα μηχανοργάνωσης κτλ. Τελευταίο σημείο. Δεν είμαστε υπουργοί για να ορίσουμε τον προπολογισμό. Έχουμε σημαντικέ προτεραιότητε. Σα παρακαλώ ένα τελευταίο σημείο για το χρονοδιάγραμμα. Συγγνώμη για το χρονοδιάγραμμα. Πέμπτη στι 12 λίγη προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών. Όσοι τον το λέω αυτό, είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Συγγνώμη, γιο, γιο, γιο πρέπει να το πω. E, ναι, θα ήθελα Θα ήθελα να μιλήσω για την τροπολογία 22. Η Φρανσουάζ μιλάει εδώ για την προτέρα έγκριση και το Συμβούλιο θεωρεί ότι η προτέρα έγκριση δεν πρέπει να χορηγείται αν ε, αυτό είναι υπέρ του γενικού συμφέροντος, ε, αν ε, μπορεί να υπάρξουν εμπόδια στη διασυνοριακή υγειονομική περιθέλψη. Αυτές οι γενικές διατυπώσεις με προβληματίζουν. Έχει τύχει να μην πάρει κάποιος διαβατήριο γιατί υπήρχαν τέτοιες γενικόλογες διατάξεις. Ας μου εξηγήσει η Φρανσουάζ. Δεν δίνεται η προηγούμενη έγκριση αν υπάρχει κίνδυνος ε, ε, αν ε, μπορεί να κινδυνεύσουν γενικότερα κοινωνικά συμφέροντα. Δηλαδή τι, τι, πώς θα κινδυνεύσουν, σε ποιες περιπτώσεις ας μπορεί η έγκριση να μην δοθεί. Εντάξει, πάλι θεωρεί... Α, η Κομισιόν, Γενική Διευθύντρια από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη Φρανσουάζ Γκροστέτ για την παρουσίασή της. Υπάρχει λόγος που είμαι εδώ. Ε, για, μας, είναι πολύ σημαντικό να παριστάμεθα σε αυτήν την πρώτη συζήτηση ούτως ώστε να, να καταλάβουμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Η πρόταση της Επιτροπής αρχικά ήταν πολύ φιλόδοξη και μας άρεσε η πρόταση ανάγνωση. Μα άρεσε το γεγονό ότι υποστηρίξατε και εσεί τη φιλοδοξία μα στα πλαίσια τη πρώτη ανάγνωση. Αλλά η διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο ήταν δύσκολη, όπω είπε η Dagmar Ροτμπέρεντ. Ήμασταν πολύ, κοντά πολύ κοντά συγγνώμη, σε αδιέξοδο. Ε, πολύ κοντά στην αδυναμία ύπαρξης κοινή θέση. Οι Υπουργοί όμω συνειδητοποίησαν ότι εδώ μιλάμε για θεμελιώδη δικαίωμα των ασθενών. Πρέπει οι ασθενεί να μπορούν να μετακινούνται και γι' αυτό οι Υπουργοί πρέπει να κάνουν κάποιε υποχωρήσει. Μιλάμε για ένα τομέα όπου τα κράτη-μέλη παίζουν το χαρτί της ε, ε, βιωσιμότητα των προπολογισμών του. Οι Υπουργοί Υγεία φυσικά έχουν κάποιες ευθύνες για να υπάρξει βιωσιμότητα του προπολογισμού, του εθνικού προπολογισμού. Εμείς λοιπόν για αυτό τον λόγο ως Κομισιόν υποστηρίξαμε την κοινή θέση που βάζει αυτό το σύστημα πρώτερη έγκριση που δεν υπήρχε στη δική μα πρόταση. Το υποστηρίξαμε για αυτό το λόγο, για λόγου δημοσιονομικού. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Και το καταλάβαμε το γιατί. Να αναφερθώ πάλι σε αυτά που είπε η Ντάκμαρ. Πρέπει να εφαρμοστεί πραγματικά, ειλικρινά και τίμια αυτό το νομοθέτημα. Θα πρέπει σε κάποιε περιπτώσει το κράτος μέλος να, μπορεί να λέει δεν δίνω αυτή την έγκριση. Γιατί αυτή η έγκριση θα είναι εις βάρος ε, της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας μου. Αυτό γίνεται για λόγους τιμιότητας, δεν γίνεται για λόγους διακρίσεων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα τα οποία επιτρέπουν σε έναν Υπουργό Υγείας να λένε Φτάνω μέχρι εδώ. Εδώ δεν μπορώ να προσπεράσω αυτό το όριο. Δεν μπορώ να πληρώσω παραπάνω. Δεν έχω τα λεφτά. Από την άλλη όμω, όταν δεν υπάρχει λόγο και δεν συντρέχει τέτοιο πρόβλημα οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα, θα πρέπει τότε ο κατάλογο των κριτηρίων να μην είναι ανοιχτό και ιστοδυναικέ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει. Εδώ μπορούν τα κρατημέλη να κάνουν προσπάθεια και να καθορίσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό κριτηρίων στα πλαίσια ενό καταλόγου κλειστού. Σε σχέση με την πρώτερη έγκριση, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει μια κίνηση, μια χειρονομία. Η κυρία Γκροστέτ θα πρέπει να κάνει μια χειρονομία για να ηρεμήσει το Συμβούλιο. Για την ε, ενημέρωση του ασθενού. Φυσικά, ο ασθενή που θέλει να μετακινηθεί, καλό είναι να ενημερώνεται. Είναι σημαντικό αυτό. Λίντα Μακέβαν, να σου πω κάποια νούμερα. Σήμερα το λιγότερο από το 1% των ασθενών μετακινούνται. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία θα αυξήσει αυτό το ποσοστό. Γιατί οι ασθενεί, όταν μπορούν να θεραπευτούν, τέλο πάντων να λάβουν αγωγή κοντά στο σπίτι του, στη χώρα του, προτιμούν να μείνουν εκεί. Αν το πολύ πολύ να γίνει 2%. Επομένω το νούμερο είναι πολύ περιορισμένο. Υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν να δίνουμε, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δίνουμε ενημέρωση στον ασθενή και πληροφορίε στον ασθενή. Επίση, ο ασθενής αυτός να μπορεί να έχει τα μέσα να μετακινηθεί. Πρέπει να υπάρχει και μια μορφή προκαταβολής βέβαια. Μια και υπάρχει αυτό το σύστημα της πρώτερης έγκρισης, τα κράτη-μέλη θα γνωρίζουν για ποια θεραπεία μιλάμε και για τι ποσά μιλάμε. Επομένως, για ορισμένε περιπτώσεις θα είναι σε θέση να επιβάλλουν μια προκαταβολή. Για τις σπάνιες ασθένειες τώρα. Αυτός ο κανονισμός μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ορισμένες σπανείς αρρώστιες. Ένα άτομο το οποίο πλήττεται πάσχει από μία σπάνια αρρώστια με βάση τον κανονισμό κοινωνικής περίθαλψης μπορεί να μετακινηθεί ζητώντα μία πάσια κόσμος δεν ξέρει τι υπάρχει αλλού. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια υποδομή για την κινητικότητα. Και με αυτόν τον κανονισμό πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη γνώση για τις ε, σπάνιες αρρώστιες. Ε, θα βελτιωθεί και η ικανότητα διάγνωσης παράλληλα. Ο Επίτροπος Άσκας ε, μας ζητάει να αξιολογήσουμε τον, το ποσοστό των σπάνιων ασθενειών και τα χρήματα τα οποία, για τα οποία μιλάμε. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε όλε τι θεραπείες, όλε τι αγωγέ για όλε τι σπάνιες αρρώστιε κάθε φορά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια βιώσιμη λύση και να βρεθεί μια ισορροπία για την ε, ηλεκτρονική υγεία. Και εμεί ε, πολεμήσαμε με το Συμβούλιο για να περάσουμε αυτό που προσπαθεί να περάσει τώρα σε τροπολογία η κυρία Γκροστέτ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, εφαρμογή των κανόνων, η ηλεκτρονική υγεία βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών, υπάρχει μια συνέχεια στη θεραπεία τους και νομίζω ότι περικόπτονται και, τα, και οι ιατρικές δαπάνες. Θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση, ούτως ώστε η Κομισιόν να συνεργάζεται περισσότερο για αυτό το θέμα με τα κράτη-μέλη, το θέμα της ηλεκτρονικής, της ηλεκτρονικής υγείας, για τα ποιοτικά κριτήρια. Τώρα, είναι σημαντικό στην οδηγία να υπάρχει μία βάση για να δουλέψουμε επί κριτηρίων ποιότητας και επί του κριτηρίου της ασφάλειας των ασθενών. Σήμερα δεν είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τέτοια κοινά κριτήρια ποιότητας. Η κατάσταση διαφέρει πολύ από κράτος μας και κράτος μέλος. Η κοινή θέση μας δίνει μια βάση. Λέει ότι απόκειται στο κράτος μέλος της θεραπείας να καθορίσει τα κριτήρια ποιότητας. Το κράτος μέλος στα πλαίσια τα δικά του αποφασίζει ποια είναι αυτά τα κριτήρια. Και το άλλο κράτος μέλος που πρέπει να επιστρέψει τα έξοδα λέει, ωραία, αν το πρώτο κράτος μέλος εφόσον το κράτος μέλος κάποια πράγματα δεν αναγνωρίζει ότι εντάσσονται μέσα στα κριτήρια ποιότητας, εγώ δεν επιστρέφω αυτά τα ιατρικά έξοδα. Φυσικά, λοιπόν, ε, για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε κοινά κριτήρια ποιότητας. Για να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα είναι θεμελιώδες. Όχι μόνο γιατί δίνει νομική βάση στους Ευρωπαίους ασθενείς για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά και γιατί δημιουργεί μια βάση για να συνεργαστούμε σε ορισμένους τομείς, ούτω ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικό σύστημα, να υπάρχει σύγκληση όπου είναι δυνατόν, να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία επίση. Κάνω έκκληση λοιπόν. Πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό και μάλιστα γρήγορα. Θα ήταν κρίμα να μπούμε σε μια διαδικασία ατέρμονης συνδιαλλαγής. Α μα βοηθήσει το Κοινοβούλιο με μια θέση που θα βοηθήσει την επίτευξη συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Okay. Thank you. Uh, Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας κομισιόν. Φρανσουάς Γκοστέτε. Εσύ έκανες μια πολύ εκτεταμένη παρουσίαση. Μάθε όμως ότι τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σου δίνω το λόγο λοιπόν για δύο λεπτά. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους Περέιρο και Εβάης Γέρπερ ότι που δεν θα μιλήσουν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δύο λεφτά η Φρανσουά και κλείνουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλους τους συναδέλφους. Ε, θέλω βέβαια πρώτον να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί όλοι έχουν επίγνωστο ότι πρέπει να προχωρήσουμε όπως και δίποτε και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι ενδιαφέρον για τους ασθενείς. Θέλω απλά να καθησυχάσω ορισμένου από του συναδέλφου που ανησυχούν ιδιαίτερα, τουλάχιστον περισσότερο από κάποιου άλλου, για τον ε, πληθωρισμό τον ε, της περίθαλψης σε κάποια κράτη-μέλη. Ακούγονται στο Συμβούλιο, ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι αφορά ένα ελάχιστο ποσοστό που είναι κάτω της μίας ποσοστίας μονάδας, κάτω του 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Και ξέρουμε ότι συνήθως προτιμούμε να Έχουμε την, την υγειονομική πέθαψη στη χώρα μας ε, και δεν θα πάμε εύκολα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε λίγο σχετικά τα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά την πρώτερη έγκριση, με αυτό το μέτρο και με την επιστροφή των δαπανών από το κράτος μέλος. Σε σχέση με το τι θα επιστρεφόταν ως έξοδο αν γινόταν στο κράτος μέλος που είναι ασφαλισμένος ασθενής η θεραπεία του, νομίζω ότι απαντώ στις ανησυχίες και στα ερωτήματα που έθεσαν ορισμένοι συνάδελφοι. Πραγματικά θέλω να σας καθησυχάσω. Άπαξ και βάλουμε κατά μέρος τα προβλήματα αυτά, διότι έχουμε τις απαντήσεις για τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε πράγματι να επεξεργαστούμε συμβιβαστικέ προτάσεις. Αν θέλουμε στη δεύτερη ανάγνωση να έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα, γιατί αυτό θα είναι καλό καλή, μια μεγάλη επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί υπάρχουν προσδοκίες. Και επαναλαμβάνω, αυτό που σας προτείνουμε είναι πραγματικά η απόρρια, η συνέπεια των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίποτα περισσότερο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που φύγει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι στις 27-28 Οκτωβρίου πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Χρειάζονται 15 ημέρες εργασίας για τις πολλές τροπολογίες που θα κατατεθούν για να γίνουν όλα όπως πρέπει. 39 του στις 6 το απόγευμα, στις 12. Ο Φάκελος είναι γνωστό εδώ και μια εβδομάδα. Η κοινή θέση είναι γνωστή από το Μάιο. Λοιπόν, 39 του στι 18 είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ για την συμμετοχή των συναδέλφων και να πω ότι τώρα με το καινούργιο εργαλείο ηλεκτρονικά, το electronic tool θα είναι ε, αυτό που θα χειριστεί τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε λοιπόν τους πάντες και την κυρία Γκροστέτ και όλους. Λύεται τη συνεδρίαση.